Bonjour à tout le monde. Nous allons commencer la réunion de notre commission par l'adoption de l'ordre du jour. Λοιπόν, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, από εκεί ξεκινάνε τις εργασίες. Τώρα, όσον αφορά τη διανεμηθήσα ημερήσια διάταξη, έχουν προταθεί δύο αλλαγέ και σα προτείνω τι δύο αλλαγέ. Πρώτη αλλαγή, τη ζήτησε η κυρία Στρίφλερ. Συμφώνησε ο κ. Πρέντα να αντιστρέψουμε τη σειρά της ανταλλαγής απόψεων των δύο συγητών. Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο ουσιαστικό σημείο με το σχέδιο γνωμοδότηση της κυρίας Τρίφλερ όσον αφορά τη συμφωνία ΦΛΕΚΤ και μετά τις δύο γνωμοδοτήσεις της κυρίας Σαρτζεντίνη και στις 16 και 5 το σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Πρέντα θα συζητήσουμε όσον αφορά την ελευτική συμφωνία με το Μαρόκο. Η κυρία Κρετού ζητάει ανταλλαγή απόψεων όσον αυτό σχέδιο γνωμοδότησή τη, όσον αφορά την σεξουαλική εκμετάλλευση και την πορνεία, να αναβληθεί για τη συνεδρίαση τη 4 και 5η Νοεμβρίου. Στη θέση αυτού του σημείου θα συζητήσουμε τι τροπολογίε όσον αφορά το σχέδιο γνωμοδότηση του κυρίου Πρέντα, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ε, που θα. Ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και μετά έχουμε και την γνωμοδότηση του κυρίου Γκούσταυσον που θα συζητηθεί γύρω στις 5 Έχετε αντιρρήσει να αφορά την τροποποιημένη τώρα ημερήσια διάταξη. Όχι, λοιπόν ε, εγκρίνεται. Λάβατε τα πρακτικά της συνεδρίασης της 16-17 Σεπτεμβρίου της Επιτροπής μας. Αν έχετε κάποιες παρατηρήσεις, τις γνωστοποιείτε στην ε, γραμματεία πριν το τέλος της ε, σημερινής συνεδριάσεως. Διαφορετικά, αν δεν υπαρβληθούν παρατηρήσεις, θα θεωρηθεί ο εγκεκριμένο το κείμενο των πρακτικών έχετε λάβει και έχετε στο φάκελό σας την ε, συστάσεις και τις αποφάσεις των συντονιστών που έγινε στις 10 Οκτωβρίου του 2013. Αν έχετε παρατηρήσει όσον αφορά τα αποτελεσμάτα της συνεδρίας των συντονιστών, να επισημάνετε τις παρατηρήσεις σας στη γραμματεία πριν το τέλος της σημερινής μας συνεδριάσεως. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, τα αποτελέσματα αυτά θα εγκριθούν όσο έχουν. Έχω μία ανακοίνωση να σας κάνω. Ήμουνα σε ένα συμπόσιο το Σάββατο από μία μη κυβερνητική οργάνωση. Βιβλιοθήκη χωρίς σύνορα είναι η ονομασία της μη κυβερνητικής οργανώσεως. Ο Πατρίκ Βέιλ τη διευθύνει και προσπαθεί αυτή να θέσει τον πολιτισμό στα πλαίσια στην έννοια της ανθρωπιστικής βοηθείας. Αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση εκλήθη στην ΑΕΤ ε, μερικές μέρες μετά την καταστροφή και υπήρχε μεγάλη ανάγκη να μοιραστούν ε, βιβλία και επεχτούνται τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες. Ήταν μια πρωτοβουλία που έγινε πολύ θετικά δεκτή. Ε, ψάξαμε να δούμε ποια ήταν η θέση του πολιτισμού στην ανθρωπιστική βοήθεια και είδαμε ότι δεν υπάρχουν ειδικέ αναφορές, διατάξεις, κονδύλια από τον προπολογισμό για να καλυφθούν οι σχετικές ανάγκες και νομίζω ότι αν κοιτάξουμε το θέμα από κοντά βλέπουμε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια περιορίζεται χρονικά σε ένα εξάμεινο αλλά πολύ συχνά τα εκτοπιστέντα άτομα περνούν πολύ μεγάλο χρόνο στα στρατόπεδά τους Μέσω 17 ε, χρόνια είναι, μπορεί να είναι η ε, παραμονή. Λοιπόν, η παιδεία και ο πολιτισμός ε, θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται και ίσως αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί και ήθελα αυτό να το μοιραστώ μαζί σας και θα το προτείνω και στους συντονιστές να διοργανώσουμε μια μικρή ανταλλαγή απόψεων με την μη κυβερνητική οργάνωση Βιβλιοθήκη Χωρίς Σύνορα ε, διότι νομίζω ότι υπόσχεται πολλά η προσπάθειά της και είναι χαμηλό το κόστος της προσπάθειας σε σχέση με τα αποτελέσματα που δίνει και την υποστήριξη που δίνει στα εκτοπιστέντα άτομα που έχουν χάσει το σπίτι τους. Η, Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της έχει μια ανακοίνωση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάποια ανακοίνωση να κάνει. Εντάξει, δίνω το λόγο στην κυρία Κατρίν Μέτεπέγγεν. Α, δεν λάβαμε ερωτήσεις για να θέσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη σημερινή, για τη σημερινή συνεδρίαση. Πάμε στην ανταλλαγή απόψεων σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Τίφλερ για την τροποποίηση του κανονισμού τη... 2173 του 2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ενός ε, σχήματος, ε, δι, ε, σχήματος αδειοδότητης FLEX όσον αφορά την εισαγωγή ξυλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα σχέδιο γνωμοδότης Επιτροπής ΙΝΤΑ που είναι καθήλυνα αρμόδια. Η νομοθετική πρόταση δεν θέλει να τροποποιήσει το περιεχόμενο του καθεστώς αδειοδοτήσεως FLEX αλλά ευθυγραμμίσει τι διατάξει τη στα πλαίσια τη επιτροπολογία. Είναι οι κανόνε που αφορούν τι κατεξοδότηση πράξη και τι εκτελεστικέ πράξει. Κυρία Στίφλερ, λοιπόν, έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε τη γνωμοδότησή σα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτή η πρόταση τη επιτροπή έχει σαν στόχο να ευθυγραμμίσει τι διατάξει της Επιτροπολογίας με τον κανονισμό FLEX στα πλαίσια των νέων, της και τη κατεξοδότηση πράξη. Αυτό ο κανονισμό του 2005 δημιουργεί ένα σύστημα διοδότησης που ονομάζεται FLECT για να καταπολεμηθεί το πρόβλημα τη παράνομη εκμετάλλευση των δασών και του σχετικού εμπορίου. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σαν στόχο όχι την τροποποίηση της φύσεως του καθεστώτος ΦΛΕΚ, αλλά να ευθυγραμμίσει τις διατάξεις επιτροπολογίας με τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα υιοθέτηση εκτελεστικών πράξεων και κατεξουσιοδότηση πράξεων. Οι εκτελεστικέ πράξει θα υιοθετηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία τη εξέταση για την αξιολόγηση των φυσταμένων μηχανισμών που έχουν σαν στόχο το να εγγυώνται την ε, νομιμότητα και την αξιόπιστη εμπνευσιμότητα της ξυλίας και των σχετικών προϊόντων που εξάγονται από τις χώρε εταίρους τις κατεξοδότησες πράξεις που θα θεθούν ώστε να τροποποιηθεί ο κατάλογος των χωρών εταίρων και των αρχών αδειοδότησης που καθορίζονται από τις ανλόγω χώρες, καθώς και τον κατάλογο ξυλίας και των διαφόρων σχετικών προϊόντων. Προτείνω δύο τροπολογίες, μία που έχει σαν στόχο να εγγυάται το ότι η διάρκεια της ανάθεσης της, της εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι απροσδιόριστη, ανοιχτή αλλά να περιορίζεται σε πενταετία αυτή η περίοδος μπορεί σιωπηρά να παραταθεί για μια παρόμοια περίοδο. Δεύτερον, η δεύτερη τροπολογία θέλει να παρατείνει κατά δίμηνο την περίοδο που ανατίθεται στο Ευρωπαϊκό για να προβάλλει αντιρρήσει όσον αφορά ένα σχέδιο κατά πράξης. πράξη. Ε, αυτά λοιπόν, αυτέ είναι οι τροπολογίε και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Κόρτες Λάστρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Στρίφλερ για το έργο το οποίο επετέλεσε. Είναι πάρα πολύ αξιόλογο αυτό το οποίο έκανε που είναι τόσο τεχνικό, τεχνοκρατικό και θα, πρέπει να πω στην συγκέντρωση θα την υποστήριξει η πολιτική μου ομάδα. Δεν ξέρω, φορέστε και τα ακουστικά για να ακούσετε. Έλεγα λοιπόν ότι τα πει πάρα πολύ καλά γιατί είναι τεχνικό και περίπλοκο το σχέδιο το θέμα, οπότε πρέπει να σας πω ότι θα την υποστηρίξει η πολιτική μας ομάδα. Επίσης, θα ήθελα να σας πω κάποια σύντομα σχόλια όσον αφορά το περιεχόμενο για την βιοπικιλότητα, για όλα αυτά τα δάση που είναι τόσο ποικιλόμορφα. Θα πρέπει να προσέξουμε γιατί όλα αυτά έχουν τεράστιες επιπτώσει κοινωνικές, οικονομικές, οπότε γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε κάποιο είδους μέτρα προστασίας της φυσικής ομορφιάς από τις όμορες χώρες, οπότε θα πρέπει το Κοινοβούλιο να συνεχίσει την πορεία του, τόσο ώστε αυτές οι συμφωνίες να συνεχίζονται και γι' αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να προστατεύσουμε το αυριανό μας ε, περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ε, Πρόεδρο, ευχαριστώ τώρα πολύ. Δίνω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία εκπροσωπεί ο κύριος Τζον Μπαζίλη. Aussi, j'ai deux noms sur ma liste, Madame Sveta Atanasova. Ε, έχουμε όμως και την κυρία Atanasova. Α, ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Τζον Μπάζιλ δεν είναι εδώ. Κάθεν Τιούνι ονομάζομαι. Και εργάζομαι στην Εκδήλωση για το Περιβάλλον. Έχω δύο παρατηρήσει όσον αφορά το σχέδιο του κειμένου. Πρώτα-πρώτα όσον αφορά αυτή την σιωπηρή παράταση δεν ε, μας νοιάζει να υπάρχει επαορίστο αυτή η ισχύ για την ε, κατανάθεση την ανάθεση των αρμοδιοτήτων γιατί το κοινοβούλιο μπορεί να πάσα στιγμή έτσι κι να ανακαλέσει και ε, δεχόμαστε τέλο πάντων αυτήν την περίοδο με σιωπηρή παράταση σιωπηρή συμφωνία. Τώρα όσον αφορά το 2 συν 4 θα ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά την, ε, το μνημόνιο κατανόησης που υπάρχει μεταξύ μας είχαμε πει ότι θα πάμε για 2 συν 2. Αλλά είπαμε ότι αυτό θα εξεταστεί περιπτωσιολογικά. Αλλά για το φλέγγο που έχουμε αυτές τις χώρες εταίρους, γιατί εν ώψη των αποφάσεων τέλο πάντων που θα ληφθούν, οι χώρες ε, του συστήματος φλέγγ ζητούν 2 συν 2. Κυρία Στίφλερ, θέλετε το λόγο για να ολοκληρώσετε. Je prends acte de, de votre... Λαμβάνομαι υπόψη την πρότασή σας. Την είχα υπόψη μου, μου φαίνεται πιο λίγο αυτό που εγώ προτείνω, αλλά τέλος πάντων θα δούμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Maintenant, notre projet d'avis. Θα δούμε τώρα το επόμενο σχέδιο κειμένου όσον αφορά την πρόσβαση αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών σε εσωτερική αγορά τη Ένωση στον τομέα δημοσίων συμβάσεων και διαδικασίε που υποστηρίζουν τι διαπραγματεύσει για την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τη Ένωση στι αγορέ δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών. Εισήγεται η κυρία Σαρτζεντίνη. Κύριε Σαντζεφίνη, έχετε το λόγο. Εντάξει, λοιπόν, πήγαν πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα, να εξακολουθώ να απαντώ. The, um, of the... Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου για την αμοιβαιότητα όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες, περί αυτού πρόκειται, Αντί να τροποποιούμε την πρόταση που είναι νομοθετική η πρόταση, προτείνω στην Επιτροπή να πούμε στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου να, στείλει, να αναπέμψει την πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί το λέω. Διότι οι δημόσιες προμήθειες αυτές καθ' δεν αποτελούν απαραίτητα εμπόριο. είναι ένας τρόπος ούτως ώστε οι κυβερνήσεις να βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους. Να τις βοηθήσουν ε, όσον αφορά τις εργασίες τους. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί βρίσκεται εκεί και αμφισβητήθηκε το Κοινοβούλιο κατά πόσο θα έπρεπε να συζητηθεί ή θα έπρεπε να αποσυρθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόθεση είναι να, αγορά, να ανοίξει η προθεση ειναι να να ανοιξει η αγορα ε, δημοσίων προμηθειών προς την ε, Κίνα και Ινδία. Αλλά ανοίγει η αγορά όμως και για όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, όχι μόνο για την Κίνα και την Ινδία. Λοιπόν, ακόμα και όλες οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να επιτρέψουν στις ευρωπαϊκές εταιρείες να μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά τους δημοσίων προμηθειών. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα. Να παράδειγμα ας δούμε τη συμφωνία για κρατικές προμήθειες του ΠΟΕ. Είναι μια συμφωνία που δεν έχει υπογραφεί από αναπτυσσόμενες χώρες. Το συζητήσαμε πρόσφατα στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Υπήρχε και άλλη μια υπογραφή στη συμφωνία του ΠΟΕ ε, που είναι η Αρμενία, που ήταν πρώην αναπτυσσόμενη χώρα. Ήθελε η Αρμενία να είναι πιο κοντά στις δυτικές αγορές, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά είναι τυπικό φαινόμενο αυτό ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες δεν προσυπογράφουν τη συμφωνία για τις δημόσιες προμήθειες του ΠΟΕ. Βλέπουμε και κάτι άλλο. Οι ευρωπαϊκοί διαγωνισμοί ανοιχτοί προς αναπτυσσόμενες χώρες, δηλαδή ευρωπαϊκές εταιρείες που θέλουν να συμμετέχουν στις αγορές των αναπτυσσομένων χωρών για δημόσιες προμήθειες διατρέχουν κίνδυνο. Δηλαδή να αντιμετωπίσουν ενισχύσεις που χορηγούν οι κυβερνήσεις. οι ευρωπαϊκέ εταιρείε χρησιμοποιούν την αναπτυξιακή βοήθεια που χρησιμοποιούμε και θέλουμε να μην έχουμε συνδεδεμένη βοήθεια που χορηγείται με αυτό το άνοιγμα των αγορών, διότι έτσι ίσω αυξάνεται η συνδεδεμένη βοήθεια. Καταλαβαίνω τι επιθυμίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήθελε να ανοίξει την κινέζικη αγορά. Ε, δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Όμω έχω πρόβλημα τη παρενέργεια που δημιουργεί αυτό και η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιείται περί αμοιβαιότητας είναι κάτι που αμφισβητώ. Βλέποντας τι γίνεται με τις δημόσιες προμήθειες εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πόσες ξένες εταιρείε έχουν πρόσβαση στην αγορά μας των δημοσίων προμηθειών, βλέπουμε ότι είναι πολύ περιορισμένα τα πράγματα. Ακόμα και από χώρα μέλος σε χώρα μέλος οι διαγωνισμοί για δημόσιες προμήθειες πολύ συχνά ε, δεν, ανα, δεν ανατίθεται σε μια ξένη εταιρεία. Το ότι ξένες εταιρείε μπορούν να έρχονται στις δικές μας αγορές δημοσίων προμηθειών, πώς να το πω, είναι θεωρητικό ζήτημα και όχι πρακτικό. Στην πράξη δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Δεν μιλάμε για αμοιβαιότητα, διότι δεν υπάρχουν ξένες εταιρείε στην αγορά μας. Άρα, γιατί να ζητάμε και το αντίστροφο και να δυσκολεύουμε το να προστατεύουν τις αγορές τους οι αναπτυσσόμενες χώρες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να επιτρέπουμε να ανατίθενται αυτά, αυτοί οι δημόσιοι διαγωνισμοί αυτά, ε, να βρίσκουν αναδόχους σε τοπικό επίπεδο. Δεν είναι νομοθεσία αυτή που ταιριάζει με τις δικές μας ιδέες της Επιτροπής Ανάπτυξης και δεν βοηθά την ανάπτυξη. Και προτείνω να πούμε στην Επιτροπή Ίντα να αναπέμψει το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επανεξέταση. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ. Κύριε Κόρτες Λάστρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έλεγε ότι ούτε εμείς είμαστε φαντών υπέρ της ρύθμισης σε αυτόν τον τομέα, αλλά θεωρούμε ότι ο κανονισμός μπορεί να έχει κάποιο είδου ε, θεμητές επιπτώσεις. Για να σας αναφέρω τα εξή. τρια τρία. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να αφήσουμε έξω τις χώρες τις λιγότερο και γίνεται το περιοριτή μνήμα ώστε την ε, στις χώρες γενικευμένων προτιμήσεως, Συντρία και στις χέβα. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει κάποια συμμετρία μεταξύ των χωρών των δικών μας και των αναπτυσσομένων χωρών. Και τρίτον είναι το να μπορέσουμε εδώ να λάβουμε υπόψη κάποια επιχειρήματα ε, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και αυτό στη βάση της εμβιότητας. Αυτά τα τρία θέλουμε να έρθουν υπόψη από το κείμενο της έκθεσης. Je donne la parole à la Commission, représentée par M. Nils. Και τώρα, ο κύριος Νίλς Σίστερ και ο κ. Αντρέ Γένσενς έχουν το λόγο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you, Madam Chair. Um, thank you. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Έχουμε κάποιες εν θερμό απαντήσεις σε σχέση με αυτό το οποίο είπε η συγκεκριμένη κυρία Σαρτζεντίνη. Πρώτα-πρώτα, σχετικά αφορά την μεταχείριση των αναπτυσσομένων χωρών, προσπαθήσαμε να είναι σαφές εδώ ότι οι λιγότερο αναπτυσσόμενες χώρες σαφώς θα εξαιρεθούν από την εντολή της πρότασης και να μην έχουν μεταχείριση σαν ε, κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Ήδη έχουν γίνει σε άλλε επιτροπέ κοινοβουλευτικέ κάποιες συζητήσει για το μέχρι πού θα φτάσει ο ορισμό, τι πόσο θα καλύπτει η έννοια αναπτυσσόμενη χώρα. Και είπε ε, η συζήτηση ότι θα πρέπει να καλυφθούν και άλλε κατηγορίε. Η συζήτηση ακόμα εξελίσσεται. Και όσο περισσότερο εξετάσει τι γίνεται με κάποιες χώρες ε, μεσαίου ή χαμηλού ΑΕΠ, θα δει κανεί ότι διαβρύνεται ο κύκλο, έχουμε και τι χώρε μπρικ ακόμα. Αλλά επίση ορισμένοι ενδυνάμει στόχοι ακόμα δεν έχουν εξαιρεθεί γιατί βέβαια δεν θα είχε κάποιο είδους ε, επιπτώσεις ε, το νομοθέτημα. Αλλά θα πρέπει να δούμε το ότι η ενεργοποίηση αυτού του μέτρου αφορούσε τις χώρες αυτές που θεωρούμε ότι συνεχώς και κατάφορα είναι έτη δυσμενών διακρίσεων κατά της Ευρώπης, κατά των ευρωπαϊκών χωρών. Όμως θα πρέπει να κατέβουμε σε κάποιον ορισμό, αλλά να μην καταλήξουμε με το να εξαιρούμε τις χώρες οι οποίες θέλαμε να καλυφθούν από την αρχική πρόταση. Κάτι άλλο το οποίο είπε η κυρία είναι το κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων για τις ΜΜΕ. Τώρα, δεν έχουμε κάποιο ειδικού κανόνες για άλλους εμπορικούς εταίρους, Υπάρχουν, αλλά όχι στην Ευρώπη. Δεν θέλουμε να υπάρχουν τέτοια μέτρα όπω ισχύει σήμερα το κοινωτικό δίκαιο. Οπότε και εμεί δεν προσπαθούμε τίποτα να αλλάξουμε. Και έτσι να δυσκολευτεί λίγο ή πολύ η συμμετοχή των ΜΜΕ. Γιατί θεωρούμε ότι είναι η ατμομηχανία αυτή τη πολιτική, κυρίω τώρα στην κρίση. Και αυτό μάλιστα ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης. Δεν υπάρχει κάποιο είδου τέτοια πρόβλεψη στην Ευρώπη, τέτοιο καθεστώς. Γι' αυτό το, του είδους το set aside. Άλλες χώρες το έχουν. Οι ΙΠΑ ας πούμε το έχουν. Αν συγκρίνετε τι ισχύει εκεί, τι ισχύει εδώ, θα καταλάβετε ότι εμείς δίνουμε περισσότερες συμβάσεις με τους διαγωνισμούς αυτούς παρά είπα με το καθεστώ του set aside που έχουν και αυτό και τελικά αμφισβητώ το κατά πόσον ε, πετύχουν το σκοπό του οι πολιτικέ τάσει. Επίση, όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι το μέτρο αυτό δεν θα καλύψει την αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτά καλύπτονται τώρα από οδηγίε, από άλλα είδου νομοθετήματα και δεν θέλουμε να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Θα μείνει η κατάσταση όσο έχει. Τέλος, όσον αφορά το αν θα ανοίξουμε ή όχι τις ευρωπαϊκές αγορές, νομίζω ότι έχουμε προείπει ότι ένα από τα πιο σοβαρά στοιχεία που προβλέπεται σε κάποια μελέτη που κάνετε εδώ στο Κοινοβούλιο αφορούσε το άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών και καταλήξατε ότι περισσότερε αλλοδαπέ εταιρείε οι οποίε λειτουργούν εδώ όσον αφορά τι δημόσιε συμβάσει λειτουργούν μέσω θηγατρικών που έχουν την έδρα τους στην Αλοδαπή. Και είναι πιο, ε, ε, πιο αναπτυγμένες οι δικές μας ε, δημόσιες συμβάσεις και αγορές. Άρα κανείς θα μπορούσε να βγει στον τάμπο συμπέρασμα όσον αφορά αυτού του είδους τις θηγατρικές στην Αλοδαπή. Οι δικές μας εταιρείε δυστυχώς δεν έχουν τις ίδιες διευκολύνσεις για να πάνε στο εξωτερικό να δώσουν τη μάχη της των, των, των δημοσίων συμβάσεων. Πάντοτε σηκώνει συζήτηση το ποιε χώρε θέλουμε να εξαιρέσουμε ή να συμπεριλάβουμε. Αλλά κάπου θα πρέπει να υπάρχει κόκκινη γραμμή γιατί πάντα υπάρχει μια ομάδα χωρών που είναι ε, οι πιο πιθανοί, οι πιο δόκιμοι στόχοι του νομοθετήματο, αν τελικά υπάρξει ένα τέτοιο νομοθετήμα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Σαργεντίνη για να δευτερολογήσει. Ευχαριστώ πολύ. Οι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε εξαιρούνται από την πρόταση. Το είπα και στον κύριο Κόρτες Λάστας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το παρατήρησα αυτό. Όταν αναφερόμαστε στις χώρες εκείνες που προσπαθούμε να έχουμε στο στόχαστρο μας, στις χώρες BRICS, Κίνα, όλος ιδιαίτερος, ο χρησιμοποιούμενος ορισμός είναι ισομένων χωρών του ΟΣΑ. Η Κίνα εξακολουθεί να εμπίπτει εκεί. Είναι σωστό? Προσυζήτηση. Όμως εξακολουθεί να θεωρείται αναπτυσσόμενη χώρα. Αν θέλετε να έχετε μηχανισμό που έχει στόχο τις χώρες BRICS, θα πρέπει να κατονομαστούν, αλλά να μην δίνετε μια πρόταση που απλώς γενικά καλύπτει όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες και αυτές που δεν θεωρούνται οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Αυτό αντιστοιχεί στον ορισμό. Παρεξηγηθήκαμε όταν αναφέρθηκα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλω να πω μικρομεσαίες επιχειρήσει προέλευση αναπτυσσόμενη χώρα. Θα πρέπει οι κυβερνήσει αυτών των χωρών να μπορεί να βοηθήσουν τι μικρομεσαίε επιχειρήσει αυτέ. Όταν αυτή η βοήθεια χορηγείται μέσω δημοσίων προμηθειών και ήθελα να προστατεύονται αυτέ από εταιρείε εκτό τη χώρα και περιοχή, περιφέρεια. Να και το βασικό πρόβλημα τώρα. Ποιο είναι. Χρησιμοποιούμε τη δημόσια προμήθεια ή την επιδίωξη αμοιβαιότητα στη δημόσια προμήθεια για να ανοίξουμε αγορές αναπτυσσομένων χωρών. Εγώ νομίζω ότι αυτές χρειάζονται και έχουν και το δικαίωμα να προστατεύουν τις αγορές τους και την αγορά δημοσίων προμηθειών και ιδιαίτερα την αγορά δημοσίων προμηθειών. Διότι αυτές είναι αγορές όπου η κυβέρνηση μπορεί να κάνει τη διαφορά και να βοηθήσει τις ντόπιε επιχειρήσεις. Τέλος, Επαναλαμβάνω αυτά που είπα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι χώρες δεν υπογράφουν τη συμφωνία του ΠΟΕ για δημόσιες προμήθειες. Δεν τους αρέσει η συμφωνία. Θέλουν να έχουν το λόγο, το δικό τους λόγο στις αγορές τους. Και τι κάνουμε εμείς, υπονομεύουμε ξανά τον ΠΟΕ. Το κάναμε και μέσω των διμερών συμφωνιών. Και εδώ ξανά υπονομεύουμε τον ΠΟΕ με μια πολιτική για τις δημόσιες προμήθειες που αφήνει εκτός τον ΠΟΕ και υποχρεώνει τις αναπτυσσόμενες χώρες να ανοίξουν τις αγορές τους για τις εταιρείες μας. Εγώ εμένω στην πρότασή μου και ελπίζω να έχω πείσει και τους ε, συναδέλφους μου γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να επενθυμίσω ότι η προθεσμία υποβολής τροπολόγιων είναι 15 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Η ψηφοφορία επισγωματήσεως της κυρίας Αργεντίνη θα γίνει στις 5 Νοεμβρίου. Έχουμε άλλο σχέδιο τη κυρίας Αργεντίνη. Στην ημερήσια διάταξή μας. για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από μεγάλες εταιρείες και ομίλους η επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή είναι η νομική. Τώρα θα λάβει το λόγο πάλι η κυρία Σαργεντίνη. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εδώ λοιπόν εγώ είμαι πολύ θετική και μάλιστα προσπαθώ να βελτιώσω την πρόταση που έχει κατατεθεί. Ήταν σπουδαία χρονιά για την διαφάνεια γιατί είχαμε την οδηγία για τους δημόσιους λογαριασμούς και ε, την ε, διαφάνεια. Αναμένουμε ακόμη την πρόταση του Επιτρόπου Ντεγκούχτ για το εμπόριο ορισμένων ορυκτών και εδώ έχουμε την μη, τη δημοσιοποίηση μάλλον μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Εγώ νομίζω ότι είναι καλό που έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και των κοινωνικών ε, στάνταρτ για να παίξουν όμως πλήρως το ρόλο τους είναι σημαντικό να υπάρχει και η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Να παίξουν τον ρόλο τη εταιρεία δηλαδή. Ας θυμηθούμε την μεγάλη τραγωδία στον υφαντουργικό τομέα του Μπαγκλαντέ. Άλλωστε πρόσφατα, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, πάλι στον Μπαγκλαντέ σημειώθηκε άλλο σοβαρό ατύχημα με 9 νεκρούς και 50 τραυματίες στην, κοντά στην Τάκα. Εμείς θέλουμε οι εταιρείε μας να λειτουργούν υπεύθυνα η πρόταση της Κομισιόν λέγει ότι θα πρέπει οι εταιρείε να περιλαμβάνουν στις εκθέσεις που υποβάλλουν τέλη θέματα κοινωνικά ε, σχέσεων με τους ε, απασχολουμένους, αντιδιαφθοράς, ε, ε, μέτρα που λαμβάνουν κατά της δωροδοκίας κλπ. Επίσης, περιγραφή των πολιτικών τους, των ε, χαρτοφυλακίων τους και των σχετικών θεμάτων. Για μας τώρα εδώ στην Επιτροπή Αναπτύξεως εγώ προτείνω ορισμένες αλλαγές και αυτές οι αλλαγές αναφέρονται πρώτα στον ορισμό του τι σημαίνει μεγάλη επιχείρηση από 500 να πάμε στους 250 απασχολουμένους και επίσης και με χαμηλότερο κύκλο εργασιών. Αυτό το κάνω για να ευθυγραμμιστώ με άλλους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που ορίζουν ήδη τι σημαίνει μεγάλη επιχείρηση και στους οποίους κανονισμούς η μεγάλη επιχείρηση νοείται ως αυτή που έχει τουλάχιστον 250 απασχολουμένους. Άλλο, άλλη σημαντική πτυχή την οποία περιλαμβάνω στο γραπτό μου είναι να εξασφαλίζεται ότι η εταιρεία υποβάλλει αναφορά για ολόκληρη την αλυσίδα προμηθειών. Στην τροπολογία 15 της ε, προτάσεώς μου και σύμφωνα με τις αρχές και του ΟΣΑ και των ΗΕ ζητώ να λαμβάνονται υπόψη όλες οι πτυχές του κινδύνου. Επομένως και η κίνδυνη που σημαίνει η εταιρεία για την κοινωνία, που αντέχεται να προκαλεί δηλαδή στην κοινωνία. Και αυτό περιλαμβάνει βέβαια και περιβαλλοντικούς κινδύνους, αλλά και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για να μην υπάρξουν παραθυράκια, όπου ίσως να εξηγούν οι ε, εταιρείε διάφορα πράγματα, αλλά να αποφεύγουν να τα δικαιολογήσουν, εγώ στην τροπολογία 17 ζητώ αιτιολογημένη εξήγηση εάν δεν ε, δημοσιοποιεί σχετικά στοιχεία. Επίσης για τις διέπουσες αρχές για τις επιχειρήσεις καθώς και τις αρχές του ΟΣΑ που είναι δύο συστήματα που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη γνώμη μου από κάθε εταιρεία. Και εγώ ενισχύω τις διατυπώσεις και αφήνω έτσι λιγότερο περιθώριο να αποφασίσουν οι ίδιες εταιρείε ποιο μηχανισμό υποβολής αναφορών θα ε, επιλέξουν οι χώρες μέλη πρέπει να ε, βεβαιωθούν ότι θα ενισχυθεί η υποχρέωση των εταιριών και οι stakeholder μπορούν να επιλέξουν διοικητικές ή δικαστικές ε, διαδικασίες για να αναγκάσουν τις εταιρείες εν τέλει, δε περιλαμβάνω υποχρέωση αναφοράς αναχώρα για κάθε εταιρεία ή όμιλο εταιρεών. Αυτό τι σημαίνει στην γνωμοδότησή μου όταν στο τέλος των διαπραγματεύσεων της οδηγίας για υποβολή λογαριασμών και διαφάνεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή ο Επίτροπος Μπαρνιέ υπενόησε ότι θα ήταν ικανοποιημένος αν περιλαμβάναμε αυτή την υποβολή αναφορών για όλες τις εταιρείες, όχι μόνο δασοκομικές, ε, εξορυκτικέ κλπ. Αυτό έγινε βέβαια μετά από την λήξη του τριμερούς διαλόγου. Αλλά εμεί εννοήσαμε ότι θα το ήθελε αυτό ο επίτροπο Μπαρνιέ, αυτό το country by country reporting για τι μη χρηματοοικονομικές πληροφορίε. Εγώ κάνω λοιπόν την πρόταση στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Αυτοί θα κρίνουν εν τέλει. Όμω εμεί για να είμαστε συνεπεί, νομίζω θα είναι σωστό να ενισχύσουμε την προσπάθεια της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων στην, ε, στον αγώνα της αυτό. Ευχαριστώ. Ο κ. Κόρτες Λάστρα. Ευχαριστώ. Ε, είμαι εγώ σχεδοσίτης, αλλά επειδή δεν μπορούσε ο κύριος Μπέρμαν που είναι και ο συγκητής να ήταν εδώ, μου ανέθεσε να μιλήσω στη θέση του. Να ευχαριστήσω λοιπόν την κυρία Σαργεντίνη για το σχέδιο της γνωμοδότησης. Ε, είναι σύντονα αυτό το οποίο λέει με τις θέσεις της δική μας ομάδας και συμφωνεί ο συνάδελφος με αυτά τα οποία προτείνεται και όσον αφορά αυτόν τον στενό ορισμό των μεγάλων εταιριών καθώς και την αξιολόγηση του κινδύνου ε, Πάντως έχει μια παρατήρηση που ήδη έχουν συζητηθεί με την συγκεντρία για τις τροπολογίες 15 και 24. Σε αυτές τις τροπολογίες λέμε για όσον αφορά το κίνδυνο για κάποια θέματα που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο, περιβαλλοντικό αντίκτυπο και ανθρώπινα δικαιώματα. Θα προτιμούσε εκεί που λέει το σοβαρός, σοβαρός να, να ανασβηστεί και να, να, να υπάρχει αντίστοιχη έκφραση με το μία ε, έννοια ευρύτερη. γιατί θεωρεί ότι παίρνει νερό, τέλο πάντων ότι, είναι πιο φλού ο χαρακτηρισμός, το, το επίθετο σοβαρό κίνδυνο. το σοβαρός. Ο κύριος το έχει τον λόγο. Ευχαριστώ και εγώ επιθυμώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την κυρία Σαρζεντίνη για την έκθεσή τη, η οποία εντάσσεται στην προσπάθεια της Επιτροπής μας να ασκήσει επιρροή επί της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε, σε ό,τι μας αφορά εμάς, αναπτυσσόμενες χώρες. Η κυρία Σαρτζεντίνη σε κάποια τροπολογία, δεν θυμάμαι σε ποια, λέει επίσης ότι πρόκειται για την βούληση να γίνει πιο αϊφόρος η παγκόσμια οικονομία. Ωραία. Εγώ δεν θα ασχοληθώ με τις τροπολογίες, αλλά πιο πολύ με το πώς μπορούμε να επηρεάσουμε την συμπεριφορά των αναπτυσσόμενων χωρών. Να απαιτούμε από τις επιχειρήσεις μας που εργάζονται στην αλλοδαπή διαφάνεια έχει καλός. Όμως πρέπει να οδηγήσουμε και τις χώρες όπου ε, δραστηριοποιούνται οι εταιρείε μας ε, να ασκήσουν την ίδια διαφάνεια. Ερώτηση λοιπόν προς την Κομισιόν και ιδίως προς την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Αν δούμε δηλαδή στην φάση αυτή των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους μας, μήπως πρέπει να το περιλάβουμε αυτό ως αξίωση απέναντι στους εταίρους μας, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να αξιώνουν την διαφάνεια. Αυτή θα πρέπει να την αξιώνουν και όχι μόνο για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, αλλά, όλες για, τις, αλλά για όλες τις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στις χώρες τους. Δεν εννοώ δεν θέλω να σας πω τώρα ποιον εννοώ περισσότερο, αλλά στην Αφρική ιδίως η Κίνα αναπτύσσεται ραγδαία. Έτσι λοιπόν εκεί θα έχουμε μία μερίδα των εταιριών οι οποίε θα υπόκειται σε υποχρώσει διαφάνεια και μία άλλη εταιρεία, ε, ίσω τι κινέζικε, μία άλλη μάλλον μερίδα που δεν θα έχουν τέτοιε υποχρώσει. Αυτό λοιπόν χρειάζεται κάποια εξορρόπηση. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα θα πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οποία εκπροσωπεί ο κ. Νικολά Μπερνία Μπάντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ εσάς κυρία μου για την παρουσίαση του θέματος και τα σχόλια. Τον Απρίλιο η Κομισιόν ενέκρινε συγκεκριμένη πρόταση που ήταν ισορροπημένη και φιλόδοξη και τότε είχαμε επιλέξει να στοχεύσουμε τις μεγάλες εταιρείες άνω των 500 απασχολουμένων στο πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Με την ιδέα ότι το καθαρό μήνυμα που θέλαμε να δώσουμε είναι ότι δεν επιβάλλουμε νέες απαιτήσεις στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Εκφράστηκαν κάποιες ανησυχίες για ορισμένες εταιρείες που θα έμπαιναν στον ορισμό με 250 απασχολούμενους αλλά δεν έχουν την περιπλοκότητα και το μέγεθος ώστε να διαθέτουν το, τα απαραίτητα ταλέντα και ικανότητες. Πάντως συνολικά θα δείτε το στοιχείο της φιλοδοξίας μέσα στην αρχιτεκτονική της πρότασης που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην διαφάνεια. Όχι μόνο λοιπόν διαφάνεια της εταιρείας αλλά και απόδοση και ανάπτυξή τους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Εμείς λάβαμε υπόψη και τις επιπτώσεις στην ενία αγορά. Αλλά θέλουμε να δείξουμε και μια ευαισθησία η οποία εκφράζεται με το κατόφλι που έχουμε επιλέξει των 500 απασχολουμένων. Αλλά θέλω να τονίσω και πάλι ότι το μέτρο φύγει 18.000 περίπου εταιρείες μεγάλος αριθμός των οποίων 2.500 περίπου είναι ήδη διαφανής. Και άρα βλέπουμε ότι πολλαπλασιάζεται επί 6 με την παρούσα πρόταση. Άρα είναι φιλόδοξη η, εταιρεία, είναι φιλόδοξη η ε, πρόταση. Αλλά αποφύγαμε ταυτόχρονα να επιβαρύνουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς θεωρούμε ότι οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες και για τις εταιρείες και για τους stakeholder και για τους μετόχους και για τις δημόσιες αρχές. Βάλαμε όμως και ένα στοιχείο ευελιξίας ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται στις περιστάσεις και στην κατάσταση που ε, ισχύει στον τομέα τους. Έχουμε προτείνει και κάποια διεθνή πλαίσια τα οποία αναγνωρίζονται ως χρήσιμα επί του παρόντος και θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο να υπάρχει αυτή η διάσταση της ευελιξίας ώστε οι επιχειρήσεις να δημοσιοποιούν πληροφορίες που να είναι όντως ενδιαφέρουσες και να άπτονται των δραστηριοτήτων τους. Τονίζω και πάλι ότι με την πρότασή μας υποβάλλουμε την αξίωση, την απέτηση αυτή για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών με το Management Report και με τα Financial Statements και Κατά τη γνώμη μας, το να αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Σας ευχαριστώ αγαπητέ κύριε. Δίνω το λόγο πάλι στην κυρία Σαρτζεντίνη για να μπορέσει να ολοκληρώσει. Θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ για την υποστήριξη από την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Κατανοώ τα σχόλια του κύριου Γκέρενς να επιτρέψουμε στις ίδιες αναπτυσσόμενες χώρες να μπορούν να ελέγξουν την συμπεριφορά των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις επικρατείες τους. Νομίζω επίσης ότι η δημοσιοποίηση μη οικονομικών πληροφοριών επιτρέπει και στους δημοσιογράφους που ασκούν έρευνα αλλά και σε μη κρατικούς οργανισμούς και άλλους παρόμοιους ενδιαφερόμενους φορείς σε, στις αναπτυσσόμενες χώρες να μπορούν να επεξεργάζονται δεδομένα από τις εκθέσεις αυτές και να κάνουν τις σχετικές εκστρατείες επιτόπου. Αυτό το non-financial reporting νομίζω ότι μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο και για όσους ασκούν την πολιτική στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ναι, νομίζω επίσης ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι χρήσιμες για τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις, αλλά όχι μόνο για αυτές. Πρέπει να γίνεται αυτό το reporting που να δημοσιοποιεί πληροφορίες οι οποίες είναι χρήσιμες και για την κοινωνία. Γι' αυτό ζήτησα να μπουν και πληροφορίες που να ξεκαθαρίζουν τον κίνδυνο και πώς ορίζεται ως κίνδυνος που ενδεχόμενα απειλεί την κοινωνία και βεβαίως σε όλη την αλυσίδα προμήθειας διότι μπορεί να υπάρχουν και κίνδυνοι σε άλλο σημείο της αλυσίδας παραγωγής. Για παράδειγμα η μεγάλη τραγωδία του Μπαγκλαντές που δεν είναι μονάχα κίνδυνος για ε, την κοινωνία αλλά και για την ίδια την επιχείρηση. Σχετικά με τον ορισμό του τι σημαίνει μεγάλη επιχείρηση, εγώ προτίμησα τον ορισμό που χρησιμοποιείται, έχει χρησιμοποιηθεί ήδη και παλαιότερα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και νομίζω ότι είναι καλό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παραμείνει συνεχτικό στα νομοθετήματα που ψηφίζει και με τα άλλα νομοθετήματα. Νομίζω ότι αύριο είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, κυρία Πρόεδρε. Ασφαλώς. Όντως η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι μέχρι αύριο στις 5 το απόγευμα. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Έκθεση του κυρίου Πρέντα για την Επιτροπή Αλίας. Σημαντική γνωμοδότηση για την Ελευτική Συμφωνία με το Μαρόκο. Ο κύριος Πρέντα απουσιάζει. Είναι καθοδόν όμως. Προτείνω να μην φύγουμε από την αίθουσα. Είναι στον ανελκυστήρα, κύριος Πρέντα. Διακόπτουμε για δύο λεπτά. Μπορεί να κάνετε κανένα τηλέφωνο το μεταξύ και μετά θα συνεχίσουμε τις εργασίες όταν θα έρθει ο κ. Πρέντα. Bien, la Commission reprend ses travaux. Monsieur... να συνεχίσουμε τις εργασίες. Ο κ. Μπρέντα είναι παρόν. Euh, Θα μας παρουσιάσει λοιπόν την γνωμοδότησή του για την ελευτική συμφωνία με το Μαρόκο. Έχετε το λόγο κύριε Μπρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας Πρόβλεπα ότι θα έπρεπε να είμαι εδώ στι 16 και 25. Μου σε συνεδρία. Λοιπόν, αφορά το πρωτόκολλο Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με το Βασίλειο του Μαρόκου που καθορίζει τι δυνατότητε αλληλευτικέ και το αντιστάθμιο το οικονομικό που προβλέπει αυτή η συμφωνία τη εταιρική σχέση την αλληλευτική συμφωνία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Βασιλείου του Μαρόκου. Η Επιτροπή Αλίας είναι καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Το σχέδιο γνωμοδοτήσεως αφορά μια συμφωνία σημαντικότατη για την Ένωση. Είναι η δεύτερη πιο σημαντική αληφτική συμφωνία που έχει συναυθεί με αναπτυσσόμενη χώρα. Μετά από αυτή που ψηφίσαμε την περασμένη εβδομάδα με τη Μαυριτανία. Λοιπόν, το, Μαυρό, το Μαρόκο έχει προνομιούχες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει συμφωνία σύνδεσης. Και υπάρχει προθυμένο καθεστώς που χορηγήθηκε εδώ και πέντε χρόνια το έτος 2008. Σημαντικότατη λοιπόν η συμφωνία για το Κοινοβούλιο στο βαθμό που διαδέχεται ένα κείμενο η έγκριση του οποίου απερίφθη το Δεκέμβριο του 2011. Το παρόν πρωτόκολλο το διαπραγματεύτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει διαπραγματευτικής εντολής που έδωσε το Συμβούλιο το Φεβρουάριο του 2012 μετά από διευρυντικές επαφές για να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ των εταίρων οι επίσημες διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2012 το κείμενο μονογραφήθηκε τον Ιούνιο πέρσι μετά από έξι γύρους διαπραγματεύσεων δυσκόλων και στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων τα βασικά σημεία ήταν τα εξή. Η οικονομική συνεισφορά που καταθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω τη Ελευθερική Συμφωνία και λαμβάνονται υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να υπογραμμίσω ότι δεν πρόκειται περί απλής επαναλήψεω του προηγουμένου κειμένου, πρόκειται περί συμφωνίας που είναι ουσιαστικά νέα και που σε μεγάλο βαθμό από τι επικρίσει που διατύπωσε το Δεκέμβριο του 2011 το Κοινοβούλιο. Υπενθυμίζω τι είχαμε τονίσει Τρία σημεία είχαμε τονίσει. Πρώτον, κόστου κόστους-οφέλους, που θεωρήθη ότι δεν ήταν πολύ καλή σχέση. Δεύτερον, έλεγαν ότι το πρωτόκολλο δεν εγγυείται την βιωσιμότητα των εκμεταλλευομένων αποθεμάτων. Και τρίτον, στις επικρίσεις αναφερόταν ότι το πρωτόκολλο δεν σεβόταν το διεθνές δίκαιο στο βαθμό που δεν απεδείκνει ότι οι ντόπιοι πληθυσμοί θα ωφελούνται από τις οικονομικές και κοινωνικές ε, συνέπειες του, των διαφόρων πρωτοκόλων των σχετικών. Όπως υπογραμμίζεται και στο σχέδιο γνωμοδοτήσης που έχετε μπροστά σας, που συνέταξα αυτά τα τρία σημεία, κατά την άποψή μου, βελτιώθηκαν και τα τρία. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τη σχέση κόστους-οφέλους αναφέρουν σε τρία σημεία που είχαμε θίξει σαν Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο του 2011. Σχέσεις κόστους ωφέλους. Αυτή η σχέση έχει βελτιωθεί αισθητά. Οι δυνατότητες οι αλληλευτικές βελτιώθηκαν. 33% σε σχέση με το πρώτερο ε, πρωτόκολλο είναι μεγαλύτερος όγκος αλλά μείωση του αριθμού των σκαφών που έχουν την άδεια να αλλιεύσουν. Από 137 πάμε στα 126 σκάφη. Υπάρχει μείωση σκαφών, αριθμού σκαφών, αλλά αύξηση κατά 33% όσον αφορά τον αλλιευόμενο όγκο. Η οικονομική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μειώθηκε από 36 σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Και δίνεται μια ενίσχυση 10 εκατομμύρια για πρόσβαση στις, στις, στις πηγές. Η οικονομική συνεισφορά της Ένωσης μειώθηκε, αλλά δώσαμε συνεισφορά στην αλευτική βιομηχανία, ύψους 10 εκατομμυρίων. για την οικονομική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ενώσης και είναι σημαντικό αυτό. Περίπου το ίμιση από τα 30 εκατομμύρια έχει προορισμό την ανάπτυξη αλίας στο Μαρόκο εφαρμόζοντας το σχέδιο αλλιετής το σχέδιο αλλιευτής. Έχουμε μια αύξηση λοιπόν, πήγαμε στα 13,5 εκατομμύρια, μικρή αύξηση. Και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για τη δική μας Επιτροπή. Όσον αφορά το δεύτερο στοιχείο, η βιωσιμότητα των εκμεταλλευομένων ε, πόρων. Η αρχή της βιωσιμότητας γίνεται σημαντική συνθήκη για τη αστεριότητα. Αναφέρεται σαφώς η αρχή αυτή στο πρωτόκολλο. Ελήφθη υπόψη στις διαπραγματεύσεις. Τα βασιζόμενη σε επιστημονικά δεδομένα, τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που αφορούν τα αποθέματα, και τις, πιθανό, τις πιθανές εξελίξεις κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής και χρησιμοποιώντας και τις δυνατότητες που προβλεπόταν όσον αφορά την Ελία στο πρώτερο πρωτόκολλο. Τα αλλιεύματα από τα ευρωπαϊκά σκάφη θα ελέγχονται περισσότερο από μικτές ε, αποστολές, από ελεγκτές επί του σκάφους και από ελέγχους ε, δορυφορικούς. Οι λεπτομέρειες ε, βρίσκονται στο κείμενο. Είναι μακροσκελές το κείμενο όσον αφορά τους ελέγχους, παρατηρητές στο σκάφο κλπ. Πολλές λεπτομέρειες αναφέρονται, ο καθένας από εμά μπορεί να τις ελέγξει. Διαβάζετε στο κείμενο. Τρίτον, οι οικονομικές κοινωνικέ συνέπειε του πρωτοκόλλου για τον ντόπιο πληθυσμό, για του ντόπιου πληθυσμού. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να αποτιμηθεί. Το Μαρόκο θα πρέπει περιοδικά να υποβάλει λεπτομερεί εκθέσει αυτό συμβιβασμό όσον αφορά τη χρήση του οικονομικού αντισταθμίζατος που διατίθεται στον τομέα, καθώς και οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες επιγεωγραφικής βάσος, προβλέπεται στο άρθρο 6 του πρωτοκόλλου αυτού. Έχετε ένα άρθρο λοιπόν, το οποίο αναφέρει σαφώς ότι το Μαρόκο πρέπει σε περιοδικά χρονικά διαστήματα να υποβάλει λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιεί η χώρα τους πόρους από την οικονομική αντιστάθμιση για τη στήριξη των τόπιων πληθυσμών. Παρόμοια ρήτρα εμφανιζόταν και στο προηγούμενο πρωτόκολλο. Η βασική διαφορά ποια είναι. Ότι υπάρχουν μεγαλύτερες απαιτήσει παρακολούθησης και εποπτείας σε τρία επίπεδα. Εκθέσεις προόδου για την εφαρμογή μεσοπρόθεσμα όσον αφορά την τομεακή στήριξη και τελική έκθεση εφαρμογής πριν την εκπνοή του πρωτοκόλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που εκπροσωπείται από τη Μικτή Επιτροπή σύμφωνα με Συμφωνία θα μπορεί να αξιολογεί με γεωγραφική βάση τις συνέπειες, τα αποτελέσματα της συμφωνίας, τον αντίκτυπο για τον τόπιο πληθυσμό. Πιστεύω ότι εδώ έχουμε σημαντικό εργαλείο. Ενισχύεται από την προοδευτικότητα και την αιρεσιμότητα της οικονομικής συνεισφοράς κάτι που είναι σαφώς καθορισμένο. Και το υπογραμμίζω αυτό. Υπάρχουν δυνατότητες, δυνατότητες βελτίωσης της ε, απασχόλησης μαροκινών αλλιών σε ευρωπαϊκά σκάφη. Υπάρχουν σαφείς αναφορές όσον αφορά τις βελτιώσεις, όλοι μπορεί να τα διαβάσουν. Έτσι μπορούμε να αποφύγουμε ιδεολογικές πολιτικές συζητήσεις που δεν αναφέρονται στους αλληλείς, αλλά σε πολιτικά προβλήματα που ε, είναι σε άλλο επίπεδο. Υπάρχουν στοιχεία λοιπόν για όλα αυτά. Μπορούμε να προσμετρήσουμε τι βελτιώσει. Τα ανθρώπινα δικαιώματα λαμβάνονται στο υπόψη στο άρθρο 1 του πρωτοκόλου. Εκεί βλέπουμε τη διατύπωση που συμφωνήσαμε σε πραγματικές. Πρέπει να ειδωθεί αυτό σε συνάρτηση με το άρθρο 8 του πρωτοκόλου που αφορά την αναστολή του πρωτοκόλλου. Υπάρχει σαφή σχέση μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμάτων του άρθρου 1 και άρθρου 8 που αφορά την αναστολή, τη διακοπή της συμφωνίας. Είναι απλούστοτο να το διαβάσει αυτός. Και σε περίπτωση παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να ανασταλεί η ισχύς. Και σε περίπτωση παραβίασης δημοκρατικών θεσμών. Είναι ένα καλό πρωτόκολλο λοιπόν που επιτρέπει να συνεχιστεί εταιρική σχέση σε ανανεωμένη βάση, ε, εταιρική σχέση μεταξύ Μαρόκου και ημών και βοηθούμε και την ανάπτυξη των τόπιων πληθυσμών συμπεριλαμβανομένου και του νότου της χώρας. Ε, με λίγα λόγια, αυτά ήθελα να πω όσον αφορά αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ο κύριος Νάισερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ βέβαια αντίθετα με τον κύριο Πρέντα βλέπω μια σειρά από πτυχές που μπορούν να επικριθούν στη συμφωνία αυτή. Πάλι λοιπόν όπως και με την παλαιότερη συμφωνία περιλαμβάνονται τα ύδατα μπροστά από τη Δυτική Σαχάρα παρόλο που δεν έχουν προηγηθεί διαπραγματεύσεις με τους Σαχράουι. Επίσης δεν υπάρχει πραγματική γνήσια ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ε, σύμβαση, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει. Υπάρχει μια συμφωνία αλίας με τη Γρυλανδία, στην οποία συμφωνία με τη Γρυλανδία υπάρχει σαφώς ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία ορίζει ότι εφόσον παραβιαστούν σημαντικές διατάξεις της σύμβασης ή των ε, διατάξεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να ανασταλεί ισχύ της συμφωνία. Το άρθρο 2 προβλέπει ωστόσο στη συμφωνία αυτή ότι με το Μαρόκο γίνονται αλλιώ τα πράγματα. Λέει ότι οφείλουν να τηρούνται οι βασικές αρχές της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων όπως περιλαμβάνονται στην ε, Παγκόσμια Διακήρυξη Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και στα αγγλικά λέει shall inspire, θα εμπνέονται από, αυτήν, από αυτό το κείμενο. Δεν υπάρχει όμως ρήτρα που να επιβάλλει κυρώσεις κατά του Μαρόκου εφόσον σημειωθούν εκεί παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ρωτώ την Κομισιόν, γιατί στη μία περίπτωση υπάρχει μια ξεκάθαρη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ στην περίπτωση της Συμφωνίας του Μαρόκου όχι. Δεύτερη ερώτηση. Η Κομισιόν έχει έρθει σε επαφή με τους πολιτικούς εκπροσώπους της Δυτικής Σαχάρας και ιδίως του κινήματος Πολυσάριο ή μόνο με τις Μαροκανικές αρχές. Τέλος, για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Δυτική Σαχάρα, μπορούμε να σας πούμε αρκετά και εγώ και ο Ιβο Βάιγκελ, διότι οι μαροκανικές αρχές μας απαγόρευσαν σε τέσσερις ευρωβουλευτές την είσοδο στη Δυτική Σαχάρα. Εγώ μπόρεσα ωστόσο να μεταβώ ένα τρίμηνο μετά και είδα πόσο απειλητική είναι η κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών οι οποίοι εκπροσωπούν του Σαχράου. Μα συνόδευαν διαρκώ αστυνομικέ δυνάμεις, ασκήθηκε μεγάλη πίεση στου ανθρώπου, του Σαχράου δηλαδή οι οποίοι ήθελαν να έρθουν σε επαφή μαζί μα, Αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα ανεχθούμε. Και για το λόγο αυτό θεωρώ ότι όπως έχει προκύψει τώρα από τις διαπραγματεύσεις η συμφωνία δεν μπορούμε να τη δεχτούμε διότι τελικώς θα είναι όλοι χαμένοι. Χαμένο θα είναι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, χαμένοι θα είναι και οι Ευρωπαίοι ψαράδες οι οποίοι θα ήθελαν να μπορούν να δραστηριοποιούνται εκεί και να, ε, αλλά υπό, υπό σωστές συνθήκες και ο τρίτος χαμένος θα είναι η Δυτική Σαχάρα. Εσείς τώρα έχετε το λόγο κύριε Βέκελ. Καλώ το κύριε Μάσνερ. Ναι, είμαι σκιώδη εισηγήτρια. Οπότε δεν έχω πρόβλημα να σα Συμφωνώ με τις ε, δηλώσεις του κ. Νόισερ. Βέβαια ο κύριος Πρέντα έχει δίκιο που λέει ότι αρχικά απορρίφθηκε η συμφωνία διότι δεν είχαν ληφθεί υπόψη επαρκώς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από την αρχή δηλαδή είχαμε πει ότι η Δυτική Σαχάρα είναι εκτός ε, μαροκάνικης κυριαρχίας, δεν μπορεί να περιληφθεί. Αυτό άλλαξε. Υπάρχουν τώρα και ορισμένα άλλα πράγματα, υπήρχαν ορισμένα άλλα πράγματα που δεν μας άρεσαν τα κέρδη δηλαδή για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την Αλία. Ωστόσο έχει επέλθει σημαντική βελτίωση. Σωστά το λέει ο κύριος Πρέντα. Είναι καλύτερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι καλύτερη η ε, προσπάθεια για την εξασφάλιση της αηφορίας, καλύτερη η χρήση των ε, κονδυλίων, αλλά βεβαίω υπάρχει πάντα το θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων που εξακολουθούν να ορίζονται πολύ αόριστα. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ πιο συγκεκριμένο. Εγώ θεωρώ ότι η ρήτρα ανθρώπινων δικαιωμάτων πρέπει να είναι αυστηρή και να μπορεί και να ελέγχεται η εφαρμογή τη και να επιβάλλονται κυρώσει. Όπω είναι τώρα το κείμενο, δεν το επιτρέπει αυτό. Γι' αυτό και πρέπει σαφέστατα, κατά τη γνώμη μου, να βελτιωθεί, όπω είπε ο κ. Νόησερ. Κατά τα λοιπά, το θέμα που τίθεται είναι ότι η Δυτική Σαχάρα δεν ανήκει στο Μαρόκο, τα ύδατα τη Δυτική Σαχάρα. Είναι διεθνή ύδατα. Επομένω, δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιο έχει πρόσβαση στα ύδατα αυτά και με τους Σαχράου δεν έχουν γίνει καθόλου διαπραγματεύσει. δεν ήταν παρόντες στις διαπραγματεύσει. Ε, το Μαρόκο δεν τους εκπροσωπεί. Να λοιπόν ένα σημαντικό σφάλμα στην διαπραγμάτευση τη συμφωνία και γι' αυτό θεωρώ ότι δεν μπορεί να ε, υπερψηφιστεί. Εκτός εάν βελτιωθεί σημαντικά η ρήτρα ανθρώπινων δικαιωμάτων και φτάσει να είναι στο επίπεδο της Γρυλανδίας. Βέβαια, είναι σωστό ότι Διεθνώ το καθεστώς της Δυτικής Σαχάρα είναι ασαφές. Δεν έχει ξεκαθαριστεί και πώς μπορούμε να κάνουμε συμφωνία λοιπόν χωρίς αυτό. Εν συνόψη λοιπόν τα ίδια ε, επιχειρήματα. Εσείς κύριε Βάγκελ. Εγώ πρόεδρε να έρθω να συμφωνήσω σε αυτά τα οποία είπαν μόλις τώρα προλύσαν τη συνάδελφοι, η κυρία Μάισνερ δηλαδή και ο κύριος Νόισερ. Επίσης, θα ήθελα να προβληματιστούμε πάνω στο πώς παρουσιάστηκε σε μας αυτή η έκθεση. South is everything what is south southern... Νο, Τι είπα να πει ότι είναι νοτιός των Βρυξελών, για τη του Μαρόκου δεν βρίσκεται η Νότια Σαχάρα, αλλά το τμήμα εκείνο του Μαρόκου που είναι στα σύνορα της χώρας. Τέλο πάντων, τι θα γίνει με το διεθνές δίκαιο. Πρόκειται για το Μαρόκο και τη Δυτική Σαχάρα. Και είναι κυρίαρχη χώρα του Μαρόκο τόσο ώστε να μπορεί να συνάψει συμφωνίες και να μπορεί να διεξαγάγει εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, οτιδήποτε είδου εμπορική επιχειρηματική δραστηριότητα. Αλλά δεν έχει το Μαρόκο το δικαίωμα, αλλά ούτε εμεί έχουμε το δικαίωμα να προβούμε σε σύναψη συμφωνιών με το Μαρόκο, οι οποίε αφορούν του πόρου φυσικού και γενικότερα ό,τι ανήκει στη Δυτική Σαχάρα που δεν είναι Μαρόκο. Τώρα να σα πω δύο λόγια όσον αφορά την ρήτρα των δικαιωμάτων. Ε, το θέμα δεν είναι η Δυτική Σαχάρα. Ξέρουμε διάφορες άλλες εκθέσεις και μελέτε που έχουν δημοσιευθεί, ξεκινώντας με το Ίδρυμα Ρομπερτ Κέννεντι, ε, αλλά και το State Department, αλλά επίσης ε, και διάφορες ε, άλλες μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οι οποίες σαφέστατα έχουν μιλήσει για την παραβίαση των δικαιωμάτων στην Δυτική Σαχάρα, αλλά επίσης και στο Μαρόκο, το οποίο έχει ιδιαίτερε κακέ επιδόσεις σε όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επομένω, θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη. Εφόσον έχουμε κάποιες συμφωνίες που αφορούν μόνο το Μαρόκο όσον αφορά τα διεθνώς σύνορα τη χώρες. Επομένω, ε, κανένα είδου ελαστικότητα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα με το Μαρόκο. Αυτό το πρωτόκολλο δεν είναι ε, κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να, θα πρέπει να προχωρήσει έτσι και θα, θα πρέπει να το αναθεωρήσουμε, πρέπει να το αναδιαπραγματευτούμε εάν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με τις βασικές αρχές μας, αλλά και με τις ε, δεσμεύσεις μας όσον αφορά το διεθνές δίκαιο και το ανθρώπινο δικαιώματα. Με a la parole. Je dois dire que c'est très frappant. Ε, θα σας πω και εγώ ότι αυτό το οποίο εντυπωσιάζει την έκθεση Πρέντα είναι ότι δεν υπάρχει καν η φράση, η έκφραση, οι λέξεις Δυτική Σαχάρα. Κάτε με. Είναι απαράδεκτο να υπογράφει ε, μια τέτοια συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία η κατάφορα παραβιάζει το Δεν γνωρίζουμε. Το τι γίνεται. με τους Σαχράουι. Ξέρουμε τι θα κάνει για το Μαρόκο. Εφόσον το Μαρόκο εκήρυξε αυτήν την αποκλειστική οικονομική ζώνη νοτίως του, του, του, πλάτου 27,4 κατά βοράν, δεν θα πρέπει εμεί να προσχωρήσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Είναι απαράδεκτο. Και επίση, η κυρία Ιζαμπελ που είναι η δεν παρίσταται στη συνεδρίαση. Όμως αυτό το οποίο σας λέω εκπροσωπούν και εκείνοι. Γι' αυτό και νομίζω τελικά θα καταφέρουμε να πείσουμε την Επιτροπή Αλίας να πει όχι σε αυτή τη συμφωνία. Και επίσης στην ε, Ολομέλεια να απορριφθεί το σχετικό κείμενο. Αυτά. Και συμπαθούμε. Αλλά το κύριο Ντέβα έχει δει στο λόγο. Uh, if he signs agreement, we are in breach of international law. Εάν επομένως αυτή η συμφωνία είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου, τότε αναγνωρίζει ε, ότι ε, είναι σε μια επικοινωνική κατάσταση και επομένως γι' αυτό και μπορεί κανείς να ε, παρέμβει εκεί. Ζουν σε σκηνές, είναι η κατάσταση τραγική. Και εμείς του έχουμε γυρίσει την πλάτη. Δέρουμε σημασία στην παραλύση των δικαιωμάτων. Εδώ πέρα πρόκειται περί νεοπικιοκρατισμού. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε εκείνου οι οποίοι δεν έχουν λέγει, ε, εκείνοι οι οποίοι δεν κρατούν τι τύχε του στα χέρια του. Και όταν πάμε παραπέρα και τους αρπάζουμε τα ψάρια για λογαριασμό μας, αυτό είναι τερατώδες θα πρέπει να πούμε στην Επιτροπή, να πάει στα κομμάτια και να επανέλθει με άλλη πρόταση. Στίφλερ, ναι, έχω μόνο δύο λέξεις να σας πω, μια που ανήκω στην ίδια πολύ με τον κύριο Πρέντα. Δεν είμαι ειδική στην Γεωργία. Ο κύριος Πόγκα ασχολείται από πλευρά μας. Όμως, σύμφωνα 100% με αυτό το οποίο είπε ο Κρίστιαν, γιατί σήμερα τα ανθρώπινα δικαιώματα είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να σταματήσουμε να χάνουμε έδαφος όσον αφορά τη μάχη εκείνη γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα να δεχθούμε αυτά τα οποία προτείνονται διότι η παραδείγμα του διεθνούς δικαίου είναι κάτι το οποίο λένε και παροξύνεται σαν φαινόμενο και να δίνουμε το πράσινο φως για τέτοια πράγματα στο όνομα του κέρδους Μάλλον πρέπει να κάτσουμε και να ξαναδούμε το θέμα. Δεν είναι δυνατόν να μην με τα ανθρωπιστικά και με την ανάπτυξη να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Είναι αδύνατο. Και ε, τώρα, να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτως ώστε να προσπαθήσουν να υπερασπιστούν αυτά τα οποία δεν σηκώνουν υπερασπιστή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ ενθαρρυντικά τα λόγια σα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή, ο οποίος συνόψισε με πάρα πολύ μέστο τρόπο το περιεχόμενο α, του πρωτοκόλλου. Υπενθυμίζω, δεν πρόκειται περί συμφωνίας, πρόκειται για πρωτόκολλο. Το 2006 ισχύει η συμφωνία. Πρόκειται για την εφαρμογή, τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας μεταξύ Βασιλείου του Μαρόκο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα στοιχεία που ανέφερε ο εισηγητής αλλά για να ευχαριστήσω και τους άλλους οι οποίοι υπέβαλαν παρατηρήσεις και ερωτήσεις έλεγα ότι όλα αυτά ετώνησαν τις διαφορές μεταξύ του πρωτοκόλλου αυτού και του άλλου το οποίο απερίφθη διότι όπως γνωρίζετε από τον Νοέμβριο του 12 άρχισαν τις διαπραγματεύσεις και από τότε ε, λαμβάνουμε συνεχώς υπόψη το ψήφισμά σας αλλά και την εντολή του Συμβουλίου. Θεωρούμε δε ότι πληρούμε τα όσα εκεί επιτάσσονται. Το του κοιτάξτε το, τι λέει το πρωτόκολλο. Να μην επιστρέψουμε πάση λεπτομέρειε, μια που τα είπε και ο εισηγητή, γιατί έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία, το οποίο τόνισε το ψήφισμα του ΕΛΚ, αλλά και το Συμβούλιο. Θα πρέπει να πιάνουν το τα χρήματά μας, βάλει φορμάνη, θα πρέπει να υπάρχει βιωσιμότητα, θα πρέπει να ε, λαμβάνουμε υπόψη την επιστημονική τεκμηρίωση ε, για την αελία κλπ. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ισχύει η των δικαιωμάτων αλλά θα ωφελούνται οι ντόπιοι ε, και ότι όλα αυτά θα ενταχθούν ξεκάθαρα ή στο πρωτόκαλο και πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα στοιχεία τα εκαλύψαμε. Τώρα, όσον αφορά το να πιάνουν ε, τόπο οι χρηματικοί πόροι, ε, ήταν δύσκολε διαπραγματεύσει, όμω, όμως, πρώτα πρώτα, εμεί ξεκάθαρα είπαμε ότι θέλουμε να προσαρμοστεί η αλληλεία ή στο ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάτι αποτελεσματικό, σε κάτι χρηστικό του υπηρεών πλευρά των μας. και βέβαια να αποφύγουμε ε, τις υπερβολικές δαπάνες, τα όσα έπρεπε να ξοδευτούν, να καταβληθούν στο τελευταίο πρωτόκολλο. Είχαμε επομένω και προκειμένου μια προσαρμογή και γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μικρότερος αριθμός αλληλευτικών σκαφών και γι' αυτό και προσαρμόσαμε και τις αλληλευτικές δυνατότητες σε σχέση με τις ε, πραγματικές μας δυνατότητες ως αλληλευτικός στόλος Έχουμε και την αντιστάθμιση, μειώθηκε κατά 17%, αντιστάθμιση αποζημίωση και όλη η πρικοδότηση ψήθηκε μόνο κατά 100% και αυτό διότι ακολουθήσαμε την βασική αρχή της νέας μεταρρύθμισης της ΚΑΠ ότι δηλαδή ε, οι αυξήσεις ε, τελικά θα ε, θα γίνουν από τους πλειοκτήτες. Αυτά έχουμε να σκέψουμε πρώτο Μαρόκο. Και γι' αυτό και η βασική αύξηση πρόκειται να γίνει από τον ιδιωτικό τομέα. Όλα αυτά, άμα τεθεί σε ισχύ αυτό το πρωτοκόλλο, όπως σας είπα, να μην αρχίσουν τώρα όλες τις λεπτομέρειες και τις τεχνοκρατικές διατάξεις, γενικά είχαμε ε, βελτιώσεις και είχαμε και ένα σώρο ε, μέτρα για να μπορέσουμε να ελέγξουμε το, τον ληφτικό στόλο αλλά επίσης είχαμε το σύστημα ε, ηλεκτρονικής αναφοράς και έτσι να έχουμε μηνιαία καταγραφή και παρακολούθηση των ηλεκτρικών δραστηριοτήτων και από πλευρά ε, κοινωνική και οικονομική. Έχουμε τι διαφορετικέ κατηγορίε, υποχρεωτικέ εκφορτώσει, landings και επίση υποχρεούνται να προσλάβουν ε, τα ελευτικά μας ντόπιου αλείς. Και γίνανε όλες αυτές οι συζητήσεις, όλες αυτές οι δράσεις ε, ε, έλαβαν ένα πλαίσιο, ένα, ένα ένδυμα βιώσιμο και αηφόρο, γιατί όλη την ώρα είχαμε συζητήσει τις δυνατότητες τις Ζητήθηκε η Συμβουλή των Επιστημόνων, μας έδωσε ένας φορέας υποπεριφερειακός, ο οποίος προσέχει τους ελευθερικούς πόρους της περιοχής εκείνης. Ακούσαμε επίσης τι μας είπε και το ερευνητικό ίδρυμα, η Ιδρύματα του Μαρόκου. Είπαμε ότι πρόκειται περί σημαντικών επιπτώσεων που θα έχουμε όσον αφορά την τομιακή στήριξη. Είπαμε να γίνει αποδέσμευση όπως γίνεται ε, σε κάθε είδους ε, διαρθρωτική αλληλευτική εταιρική συμφωνία SFPA και είπαμε ότι θα ωφεληθούν όλες οι περιφέρειες του Μαρόκου. Επίσης, έχουμε εδώ ενσωματώσει κάποιες καινούργιες αρχές που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Δηλαδή, δούμε πώς θα υπάρχει ισομερής γεωγραφική κατανομή των ωφελιών τη συμφωνία. Για κοιτάξτε τι λέει το άρθρο 6 εδώ. Και έπρεπε να συμφωνήσουμε με του Μαρόκου για το τομεακή στήριξη. Αλλά έχουμε εδώ πέρα τι σχετικέ ε, εκθέσει που υποβάλλονται σε τρία επίπεδα. Την Κοινή Επιτροπή που είναι ο φορέας ο οποίο παρακολουθεί την ε, εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Επομένω, έχουμε τώρα μια τέτοια πρώτη έκθεση πρόοδου ε, όσον αφορά όλα αυτά τα οποία συμφωνήσαμε και επίσης ε, αυτό αφορά τα ατομικά ε, ε, προγράμματα. Και μόνο λοιπόν εμείς θα πληρώσουμε άπαξ και γίνουν όσα προβλέπονται. Μόνο επομένως από τη βάση της εφαρμογή η οποία θα πρέπει να γίνεται ε, με βάση την ισομερή κατανομή και επί τη βάση του προγραμματισμού που έχουμε καταρχήν συμφωνήσει με το Μαρόκο και έχουμε μετά και κάποιο δεύτερο επίπεδο ε, αναφορών, εκθέσεων. Κάθε φορά που έχουμε ολοκλήρωση ε, κάποιο τέτοιο project, θα έχουμε μια έκθεση που θα αφορά την ολοκλήρωση και την εφαρμογή αυτή τη ολοκλήρωση του προγράμματο. Οπότε εμεί να μπορούμε να δούμε κατά πόσον η τελική ωφέλη προγράμματο αντιστοιχεί με τον αρχικό προγραμματισμό. Και επίση στο τέλο του προγράμματο θα έχουμε μια τρίτη αναφορά, έκθεση που θα είναι η τελική και η οποία βεβαίως πρόκειται να σας κοινοποιηθεί και σας και στα άλλα θεσμικά όργανα και έτσι εκεί θα μπορούμε να ε, συνοψίσουμε το τι έγινε από το πρόγραμμα και έτσι μπορούν να παρακολουθούν τα θεσμικά όργανα το τι γίνεται να δείτε ποια είναι η κοινωνική ωφέλεια Είπαμε για την κατανομή της ωφελία, των κερδών τους είπε. Και επίσης έχουν και το αρθρό 1 που τα λέει όλα αυτά και κάτι άλλο πρέπει να κλείσω, πρόκειται για κάτι το οποίο θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη και σε σχέση με το αρθρό 8. Και σας διαβεβαιώνω ότι έχουμε την νομική δυνατότητα να αναστείλουμε μονομερό το πρωτόκολλο εάν από πλευράς θεσμικών ε, ε δικαιωμάτων έχουμε παραβίαση. Πρόεδρε, σύνομαι που μακρηγόρησα, αλλά κύριε με ότι λέει το ψήφισμά σα, αλλά και η εντολή του Συμβουλίου. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Και τώρα, δύο βουλευτέ έχουν ζητήσει το λόγο. Θα δώσουμε το λόγο εις τον κύριο Νόισερ. Ευχαριστώ και πάλι κυρία Πρόεδρε. Σύντομες ερωτήσεις. Αφενός ένα σχόλιο. Μου φαίνεται ότι προδίδει με την διατύπωση της προθέσης της η Επιτροπή, η Κομισιόν δηλαδή, λέει για όλες τις περιοχές του Μαρόκου. Μαρόκου. Υπάρχουν περιοχές του Μαρόκου και υπάρχει και η Δυτική Σαχάρα. Θα πρέπει από την άποψη του διεθνούς δικαίου να χρησιμοποιεί η Κομισιόν την καθαρή νόμιμη διατύπωση. Μαρόκο και κατεχόμενα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας. Όχι όλες τις περιοχές του Μαρόκου. Δεύτερη ερώτηση. Από πλευρά της Κομισιόν διεξήχθησαν ε, συζητήσεις με το Πολυσάριο που είναι η πολιτική εκπροσώπηση του, της Δικής Σαχάρας. Τρίτο, γιατί υπάρχουν διαφορετικές ρήτρε που θεσπίζει η ε, Κομισιόν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βλέπει Γρυλανδία και Μαρόκο. Και τρίτο ή τέταρτο, έγινε αξιολόγηση το, της κατάστασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων επιτόπου στην Δυτική Σαχάρα από την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ και να Ο κύριος Ντέβα έχει το λόγο. Να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπέροχη προσπάθεια για να καλύψει τα διάφορα προβλήματα. Ερώτηση. Αν μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη. Τα χρήματα που θα δώσουμε στους Μαροκινούς θα προστατευτούν ούτως ώστε να διτεθούν και στους κατοίκους Δυτικής Σαχάρας και τι ποσοστό από τους πόρους θα τεθούν στην ε, κυβέρνηση θα διατεθεί στους πληθυσμούς της Δυτικής Σαχάρας που ζουν σε φρικιαστικές συνθήκες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στο μέτρο του δυνατού Πράγματι είναι δύσκολο και ευαίσθητο αυτό το ζήτημα. Από πλευράς πολιτικής. Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα μέσω του πρωτοκόλου. Θέλαμε να εξασφαλίσουμε το εξή. Να καλύψουμε τα σημεία που έθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2011. Απαντώ στην τελευταία ερώτηση εδώ θέλαμε να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξει γεωγραφική κατανομή. Δεν μιλάμε για ποσοστά. Έχουμε λόγο. Αν κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού στην πρώτη φάση μας δώσουν κάτι απαράδεκτο, π.χ. να χρησιμοποιήσουν την τομεακή υποστήριξη για την Ταγκέρη, την περιοχή της Ταγκέρης, θα πούμε όχι. Δεν το δεχόμαστε. Δεν ταιριάζει με αυτά που διαπραγματευτήκαμε. Πρέπει να υπάρχει σαφής γεωγραφική κατανομή σε όλες τις περιφέρειες που καλύπτονται. Αυτό μπορούμε να κάνουμε στη Μεκτή Επιτροπή. Αν μιλήσαμε σε εκπροσώπου στον Σαχράουι, αρκετές φορές τους συναντήσαμε. Δεν είναι ότι τους αγνοήσαμε. Υπάρχει θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσης Δυτική Σαχάρα. Η DG Mare υποστηρίζει τη γενική θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Τα ξέρετε καλύτερα από εμάς τα θέματα αυτά πολιτικής χρειάς. Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό που θα επιτρέπει στο θεσμικό όργανο να λάβει τα αναγκαία μέτρα για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αρκούν αυτά, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Πρέντα έχει ξανά το λόγο για να ολοκληρωθεί το θέμα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε πόρα που έχω από το να ισχυριστώ ότι μπορώ να ολοκληρώσω εδώ αυτή τη συζήτηση. Σαφείς οι θέσεις. Εκτιμώ τις διαπραγματεύσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πήρα το κείμενο του πρωτοκόλου. Το έφερα μαζί μου. Έχουμε 17 σελίδες περίπου παράρτημα. Πριν τις προδιαγραφές και λοιπά, με όλες λεπτομέρειες. Δεν συζητήσαμε τις λεπτομέρειες του πρωτοκόλου. Απογοητεύομαι όμως. Διότι ήμουν προετοιμασμένος να σας διαβάσω κάποια σαφή τμήματα του κειμένου για συγκεκριμένα μέτρα και προβλέψεις. Δεν συζητούμε όμως το πρωτόκολλο. Το προέβλεπα, λέγοντας αυτά που είπα στην αρχή. Είναι θέμα σαφούς πολιτικής επιλογής. Κύριε Βάγκελ, όταν λέτε τι είναι νότος, ξέρετε πολύ καλά τι είναι ο νότος. Το Μαρόκο αποκαλεί το τμήμα που αποκαλείται Δυτική Σαχάρα το αποκαλεί νότιες επαρχίες. Στο κείμενό μας δεν μιλάμε για νότιες επαρχίες αλλά για το γεωγραφικό νότο. Υπάρχει πάντα γεωγραφικός νότος. Δεν εξαφανίστηκε ο γεωγραφικός νότος. Διάλογος εκτός μικροφώνου. Δεν τον ακούνε οι διερμηνείς. Πρέπει να χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο, λέει σωστά η πρόεδρος. Να μιλάτε με το μικρόφωνο ανοιχτό, αν θέλετε να σας μεταφράζουν. Εντάξει, το καταλάβαμε, λέει η πρόεδρος. Μετά χαράς. Ο, βλέπω ότι η Σαβέλα Λεβίν κατέφθασε, η εμπειρογνώμων μας. Θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Πρέντα, γιατί δεν ολοκλήρωσε. θα μπορούσα να αναπτύξω μια ολόκληρη επιχειρηματολογία. Όπως αναφέρθηκε και εδώ, δυστυχώς, δεν είναι σαν να βρισκόμαστε εκτός των πλαισίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καθένας από εμά έχει άποψη. Δεν πρέπει να στιγματίζουμε εκείνους που δεν θέλουν να πολεμήσουν τις απόψεις των άλλων. Έχουμε ένα πρωτόκολλο, το διαπραγματεύτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έγινε διαπραγμάτευση με τους Μαροκινούς. Εγώ έκανα αξιολόγηση, την παρουσίασα. Βάσει σημείων που παρουσιάσαμε εμείς εδώ και δύο χρόνια. Έγιναν βελτιώσεις επί των σημείων που είχαμε θίξει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διαπραγματεύσεις ε, σημείωσε προόδους που θεωρώ σημαντικές. Εξήγησα ποιες. Δεν μπορώ να αγνοήσω το ότι να αρνηθούμε χρηματικούς πόρους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη του Μαρόκου είναι η σωστή προσέγγιση, η λογική. Αν αρνηθούμε το πρωτόκολλο, δεν θα προχωρήσει το θέμα της αναπτύξεως του Μαρόκου. Αυτό είναι σαφές. Και αν οι Ευρωπαίοι αλληλείς αρνηθούν την αλληλία στους Μαροκινούς θα το κάνουν άλλοι. και δεν ξέρω αν θα είναι τόσο προσεκτικοί τα ανθρώπινα δικαιώματα οι άλλοι. Ξέρετε ότι αυτό ισχύει. Ο μηχανισμός που αναφέρεται στο πρωτόκολλο τώρα. Να υπάρχει περιοδική παρακολούθηση και εποπτεία. Να γίνεται ανάλυση όσον αφορά την χρήση των οικονομικών συνεισφορών για την ανάπτυξη των διαφορών κοινοτήτων. Αυτός ο μηχανισμός είναι καλός. και πρέπει να έχουμε την εμπιστοσύνη ότι θα χρησιμοποιηθεί. Προσωπικά έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις διαπραγματεύσεις της, αυτή είναι η άποψή μου και πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και τις απόψεις των άλλων επιτροπών του Κοινοβουλίου. Κλείνω λέγοντας ότι δεν μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα της Δυτικής Σαχάρας μπλοκάροντας ένα πρωτόκολλο. Αλίας με το Μαρόκο. Το λέω ειλικρινά. Αν θέλουμε να σκεφτούμε το θέμα πλευράς αναπτυξιακής, πιστεύω ότι αυτό το πρωτόκολλο είναι πολύ πιο ενδιαφέρον αυτό που είχαμε για να βοηθήσουμε τους πληθυσμούς του Μαρόκου για την ανάπτυξή τους. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν μπορεί να αλλάξετε επικαλούμενη αυτή τη μάχη για τη Δυτική Σαχάρα κλπ πρέπει να συζητήσουμε το πρωτόκολλο. Αν θέλετε να μπούμε σε κατά σημείο συζήτηση και να δούμε ποιε είναι οι απόψει, να δούμε πώ μπορούμε να οργανωθούμε για κάτι τέτοιο. Αυτά και ευχαριστώ. Η κυρία Σαμπέλα Λεβίν έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με επιτρέπετε να μιλήσω εκ μέρους των, της ομάδας των Πρασίνων. Συγγνώμη που κατέφθασα αργά. Δεν άκουσα όλη τη συζήτηση. Θέλω να εκφράσω τη δική μου άποψη και την άποψη των πρασίνων. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά το πρωτόκολλο. Ήμουν εισηγήτρια για την εξωτερική διάσταση της μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Καταφέραμε να πετύχουμε πολύ ουσιαστικές βελτιώσεις βελτιώσει όσον αφορά τις συμφωνίες με τίτες χώρες και τι μορφή θα έπρεπε να έχουν στο μέλλον. Και δεν νομίζω ότι το συγκεκριμένο νέο πρωτόκολλο είναι ένα παράδειγμα πάνω στο οποίο είχαμε συμφωνήσει. Ένας ακρογωνίος λήθος των νέων συμφωνιών που πρέπει να είναι βιώσιμες είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το συμφώνησε το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο. Και η εντολή του Συμβουλίου όταν εκδόθηκε για να διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο πρωτόκολλο με το Μαρόκο ήταν ότι πρέπει να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να υπάρχει ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο νέο πρωτόκολλο. Βλέπω ότι ο εισηγητής θεωρεί ότι υπάρχει ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εν λόγω πρωτόκολλο. Φοβούμαι όμως ότι δεν συμφωνώ. Αν δείτε όλες τις άλλες συμφωνίες που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν το Μέκε Πρίνσιπε, Μαδαγασκάρι, Γρυλανδία, και κλπ. Πάντα υπάρχει πολύ συγκεκριμένη ρήτρα εκεί που αναφέρεται σε αναστολή της εφαρμογής του πρωτοκόλου και μπορεί να ανασταλεί αυτό από ένα από τα μέρη αν ένα από τα μέρη παραβιάσει ένα από τα βασικά και θεμελιώδη στοιχεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 9 της Συμφωνίας Κοτονού ή όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σαφέστατη παράγραφος σε όλα τα πρωτόκολλα εκτός από αυτό. Σε αυτό βλέπουμε μία μνήμα τη Συμφωνίας Γειτονίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως Μαρόκου αναφέρεται στην καθολική διακήρυξη ανθρώπινα δικαιώματα που θα πρέπει να διαπνέει τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της κοινότητας απέναντι στο Μαρόκο. Δεν πλησιάζει καν αυτό στη διατύπωση πέρι ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως είναι σε άλλες συμφωνίες. Και για να τονίσω ότι δεν είναι τυχαίο δεν συνέβη αυτό διότι κάποιος δεν το σκέφτηκε. Ξέρω ότι η Επίτροπος κάθε φορά ερχόταν στην Επιτροπή Αλίας και απαντούσε σε ερωτήσεις μας για τις διαπραγματεύσεις, πώς πηγαίνουν διαπραγματεύσεις για την νέα συμφωνία με το Μαρόκο και τίθεντο δύο ζητήματα. Το ένα ήταν οικονομικό και το άλλο αφορούσε τη ρήτρα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Μαρόκο είχε αρνηθεί να συμπεριλάβει μια ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη μορφή που έχουν συμπεριληφθεί τέτοιες μνήες σε άλλες συμφωνίες. Και ρήτρα αναστολής στο πρωτόκολλο αναφέρεται μόνο στην περίπτωση διαφοράς για κάτι. Δεν αναφέρεται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι δεν σέβεται αυτά που έχουν συμφωνήσει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν νομίζω ότι είναι σύμπτωση το ότι το Μαρόκο δεν ήθελε να συμπεριλάβει τέτοια ρήτρα. Μπορούμε να διαρωτηθούμε γιατί. Είναι προφανές πιστεύω. Για τον ίδιο λόγο για τον οποίο ο Ιβο Βάγκελ και εγώ και ο Βίλε Μάιερ δεν μπορέσαμε να μπούμε στο Μαρόκο όταν θέλαμε να πάμε εκεί και να επισκεφτούμε τι νότιε επαρχιέ εδάφη, αποκαλέστε τα όπως θέλετε, τις, ε, τα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας όπου είχαμε έρθει σε επαφή και με την πρεσβεία του Μαρόκου. Ήμασταν πρόθυμοι να συναντηθούμε με τον κυβερνήτη της επαρχίας και με προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέλαμε να δούμε με τα μάτια μας την κατάσταση. Δεν μας επετράπει να εισέλθουμε. Ο Ήβο και εγώ είμαστε πολύ γνωστοί ε, είμαστε πράκτορες και προβοκάτορες. Έτσι μας είπαν. Γιατί. Γιατί δεν μας άφησαν να μπούμε. Και γιατί το Μαρόκο ε, έφτιαξε τείχο μήκους 2.700 χιλιόμετρων στην έρημο διαχωρίζοντας τις απελευθερωμένες από τις κατεχόμενες περιοχές της Δυτικής Σαχάρας. Γιατί? Διότι δεν είναι δημοκρατική χώρα. Οι λαοί της Δυτικής Αχάρας δεν μπόρεσαν να τοποθετηθούν, δεν μπόρεσαν να εκφράσουν τις επιθυμίες τους για το μέλλον και την αυτοδιάθεσή τους. Και κλείνοντας, εντάχει, θα ήθελα να ενημερώσω την Επιτροπή ότι η Επιτροπή Αλίας ζήτησε νομική γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας μας σχετικά με την νομιμότητα τη αγορά δικαιωμάτων αλληλευτικών πλευρά Ευρωπαϊκή Ενώσεω στην οικονομική ζώνη τη Δυτική Σαχάρα. Διότι το Μαρόκο, από ό,τι γνωρίζω, ποτέ δεν ε, αξίωσε να ελέγχει τα, την οικονομική ζώνη των χωρικών υδάτων Δυτικής Σαχάρας. Νομίζω ότι η νομική υπηρεσία θα τοποθετηθεί και θα πει ότι πρόκειται περί διεθνών υδάτων. Αυτό έχει πολύ σοβαρές συνέπειες όχι μόνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά ποιο είναι το καθεστώς αυτών των υδάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαπραγματευτεί για αυτά τα ύδατα και να αγοράσει ελευτικά δικαιώματα σε αυτά τα ύδατα. Βασικά, εγώ θα συνέστηνα να απορριφθεί το νέο πρωτόκολλο, δεν ευθυγραμμίζεται κατά την άποψή μου με τις δημοκρατικές αρχές, θα πρέπει να το απορρίψουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξαναδίνω το λόγο στον κύριο Πρέντα αν επιθυμεί να σχολιάσει αυτά που μας είπε η κυρία Λεβίν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταλαβαίνω την άποψη της κυρίας Λεβίν. Είχε ήδη εκφραστεί σε πρώτερες συνεδριάσεις. Λυπούμε διότι δεν μπορέσαμε να λάβουμε υπόψη όλες τις πτυχές της νέας καταστάσεως που συνδέεται με τις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το μόνο μπορώ να κάνω για να ολοκληρωθεί η συζήτηση είναι να σας παραθέσω το άρθρο 1 του πρωτοκόλου, να σας διαβάσω που λέει και παραθέτω στη δεύτερη παράγραφο εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 1 της Συμφωνίας Σύνδεσης που αφορά την ανάπτυξη διαλόγου και συνεργασίας και το άρθρο 2 της ίδιας Συμφωνίας που αφορά το σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το άρθρο 2 αν επιτρέπετε θα το διαβάσω, ο σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και θεμελιδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπω αναφέρονται στην καθηγητική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμπνέει την εσωτερική και διεθνή πολιτική τη κοινότητα και του Μαρόκου και αποτελεί ουσιαστικό ε, στοιχείο τη παρού συμφωνία. Σα διάβασα αυτά. Δεν μπορώ να κάνω περισσότερα από αυτά που έκανε στην πραγματεύση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δεν μπορεί να ζητήσετε από τον συγκητή να κάνει περισσότερα. Επαναλαμβάνω αυτά που ήδη είπα προελίγου, ότι θεωρώ ότι οι διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όνομα, εν ονόματί μας αποτελούν οι διαπραγματεύσεις σημαντική πρόοδο σχέση με το 2011 και το άρθρο 1 και το 8 του πρωτοκόλου προβλέπουν μηχανισμό επαρκή όσον αφορά τον έλεγχο και την παρακολούθηση βάση της πραγματικής καταστάσεως Καταλαβαίνετε ότι έχετε αντίθετη άποψη. Εκεί είμαστε. Μέσω ψηφοφορία θα τοποθετηθούμε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή αυτό είναι. Ευχαριστώ απείρω. Ευχαριστώ πολύ. Να σα υπενθυμίσω ότι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών είναι 16 Οκτωβρίου στι 12 το μεσημέρι. Θα περάσουμε στη δεύτερη γνωμοδότηση για την οποία είναι υπεύθυνο ο κύριος Πρέντα και συντάκτης και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και εγγυήσει της ε, Ένωσης για τις Επενδύσεις μετά την απόφαση των συντονιστών της Επιτροπής Ανάπτυξης να γίνει ανταλλαγή απόψεων αφορά τις τροπολογίες που αφορούν την έκθεση θα προβούμε σε μια σύντομη συζήτηση επί των τροπολογιών που αφορούν το κείμενο του κυρίου Πρέντα για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Κύριε Πρέντα, λοιπόν, έχετε το λόγο για να σχολιάσετε τις τροπολογίες και να εξηγήσετε και τη θέση σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να μην είμαι τόσο απονομένος όσο πριν τροπολογώ ξανά να παίρνω το λόγο. Πρώτα-πρώτα θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος διότι έχουμε την δυνατότητα να μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις σε σχέση με τις τροπολογίες για την εκθεσή μου. Και έχουμε κάποιες από την Επιτροπή και άλλες 20 περίπου από συναδέλφους. Για αυτές τις 20 που κατέθεσαν οι συνάδελφοι, οι πράσινοι, από τον κύριο Στάς, και εσείς κυρία Πρόεδρε, αλλά και η κυρία Κρέσ. 13 και ο άλλος 13 και ο κύριος Ντέβα 2 για την ΕΣΥΑΡ. Γενικώ, όταν σας τονίσω ότι ένα μεγάλο τμήμα των τροπολογιών κατατείνουν να μας αποδείξουν ότι έχουμε σύγκληση απόψεων όσον αφορά τι δραστηριότητε τη ΕΤΕ, όσον αφορά τι τρίτες χώρες ε, σε σχέση με τις εγγύσει της Ένωσης. Αλλά έχουν τροπολογίες συμβαστικές. έξι συμβαστικέ πέντε με του πρασίνου και μία συμβαστική τροπολογία με του συντηρητικού μεταρρυθμιστέ. Επίση, θα πρέπει να σα πω δύο λόγια για αυτέ τι συμβαστικέ τροπολογίε και παρακαλώ να τι επιψηφίσετε όταν έρθει η ώρα γιατί νομίζω ότι είναι λογική αυτή η συμβασμή και νομίζω ότι βελτιώνουν πραγματικά την πρόταση τη ε, Επιτροπής. Γι' αυτό και νομίζω ότι όσον αφορά την χρηματοδότηση ε, μέσω των ενδιαμέσων. Η πρώτη ε, συμβαστική λέει ότι θα χρειάζεται περισσότερη ε, διαφάνεια για αυτές τις δραστηριότητες με τους ενδιάμεσους. Γιατί αυτά τα δάνεια έχουν ξεκάθαρη σε επιδράσει όσον την ανάπτυξη. Και επίσης τα δάνεια της ΕΤΕ θα πρέπει να βοηθήσουν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στις χώρες που είναι δικαιούχοι ανάλογα με τι προτεραιότητε τη εν λόγω χώρα. Η δεύτερη τροπολογία τονίζει ότι θα πρέπει η τράπεζα να, ε, συνεργάζεται με εκείνους τους ενδιάμεσου που έχουν καλό όνομα. Και πρέπει να υποστηρίζονται οι σχετικέ τράπεζε τη χώρα. Ε, τρίτον, λέω ότι θα πρέπει να προσέξουμε τα θέματα υγείας και παιδείας και επίσης θα πρέπει να προτιμούνται τα δάνεια τα οποία δίνουν προθέμενη αξία. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται εις βάρος των μακρόπνων στόχων της πολιτικής ανάπτυξης. Οι τροπολογίες 4 και 5 αφορούν το συνδυασμό των δανείων. Σημαντικό στοιχείο νομίζω γιατί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτό, το, αυτή η ανάμειξη, το συνδυασμός θα πρέπει να βοηθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη πραγματικά. Θα πρέπει να ζυγίζεται αυτός ο αντίκτυπος και άρα από εδώ είναι ευκαιρία να το υπενθυμίσουμε. Επίσης θα πρέπει να προσέχουμε για την υλοποίηση από την τράπεζα και από άλλες, άλλες θεσμικές αρχές, άλλες θεσμικά όργανα. Οπότε εδώ σε αυτό το συνδυασμό θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες στόχο. Δηλαδή είναι εδώ να έχουμε αποτελεσματικότητα και διαφάνεια. Η έκτη τροπολογία εξκαθεί το ζήτημα της υποστήριξης της τράπεζας της ΜΜΕ. Γιατί εδώ αυτό το οποίο θέλουμε είναι οι χρηματοδοτήσει να βοηθήσουν τον ιδιωτικό τομέα στις δικαιούχες χώρες. Ακόμα και αν οι σχετικές επενδύσεις από αλλού δεν πρέπει να αποκλείονται. Έχω και κάποιες προφορικές τροπολογίες. Έξι. Να βελτιώσουμε κάποιες διατυπώσεις των αρχικών τροπολογιών για την πρόταση της Επιτροπής. Παρακαλώ να εγκρίνετε και αυτές τις προφορικές τροπολογίες. καλός να σκέψη, το έκανα και πίεση χρόνου. Οπότε γι' αυτό και χρειαζόντουσαν αυτέ οι βελτίωσει. Η προφορική υπαρτιμόν 1 λέει να μην έχουμε κριτήρια επιλεξιμότητα για την χρηματοδότηση, για την απόφαση που αφορά την εξωτερική εντολή της τράπεζας. Και τη αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην βαρύνει η διαδικασία αποφασίσεων θα πρέπει αυτά τα κριτήρια να είναι προσβάσιμα από όλους. Επίσης, επισηρώ την προσοχή σας σε μια τροπολογία την οποία κατέβασα την υπόλοιπη 39. Μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα πρέπει όχι μόνο να ε, επιβάλλουμε μόνο κάποια απαιτήσει τράπεζα, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε το business model της ε, τράπεζας και να αξιοποιούνται τα όσα θέλουμε να κάνουμε την εξωτερική μας πολιτική ως Ένωση. Επίσης, θέλω να πω μπράβο στον κύριο Καλφίν, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι εγγύσεις. Voilà, donc euh, en gros c'était ce que j'ai voulu euh, vous dire euh, en guise d'introduction pour notre... Αυτά προσαγωγικά για την ανταλλαγή από... Euh, de nouveau, Euh, merci euh, de votre attention. Τώρα υποφαινομένη θα λάβει το λόγο, λέει ο Πρόεδρο, ε, για τους πρασίνους. Ε, εμεί θεωρούμε πάρα πολύ θετική αυτή η προσπάθεια για του συμβιβασμού που έκλεισε ο εισηγητή. Αυτό θέλουμε και εμεί και σα ε, τονίζω επίση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η ενδιάμεση να αποτελεί σε κάποια κριτήρια κεραιότητο και έτσι να έχουμε διαφάνεια, καταπολέμηση διαφάνειας και να βοηθάει το περιβάλλον αυτά. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βοηθούμε τις αναπτυσσόμενες χώρες και τοπικά. Αυτό είναι η έκτη τροπολογία. Επίσης, με μεγάλη μας ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι η τροπολογία 5 καλύπτει η δική μας τροπολογία όσον αφορά την αξιολόγηση του συστήματος το σύστημα αυτό της ανάμειξης δωρεών και δανείων. Και έτσι να υπάρχει συμπληρωματικότητα χρηματοδοτική. Και το σύστημα αυτό να έχει κάποιες απτές συνέπειες πάνω στη βιώσιμη ανάπτυξη. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να μην το ξεχνούμε τώρα όσον αφορά ότι θα πρέπει να τηρείται η υπευθυνότητα των αναπτυσσομένων χωρών. Η κατά τη της δικής μας ομάδας είναι πάρα πολύ προφανές ότι όλες οι επενδύσεις της ΕΤΕ θα πρέπει να φυγραμμίσουν με την στρατηγική ανάπτυξη που υπάρχει σαν εθνική πολιτική. Πρώτη είναι το πρωί 28. Οπότε γι' αυτό σας λέω ότι είναι πάρα πολύ αρνητικό το ότι το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 33 είναι διάταξη την οποία δεν θέλει ο εισηγητής γιατί θα θέλουμε αυτά τα προγράμματα μικρής κλίμακα, τα αποκεντρωμένα για την με συνέργειας που θεωρούμε ότι αυτό είναι μια καλή εναλλακτική για να μην έχουμε αρνητικές επιπτώσεις κοινωνικές και περιβαλλοντικές όσον αφορά τις, τις, τις ε, μεγάλες κλίμακας ε, υποδομές γιατί μας φαίνεται εξίσου σημαντικό ότι θα πρέπει να δούμε εδώ ότι υπάρχει μια συνέπεια το, η τροπολογία 43 όσον αφορά την μετάδοση των πληροφοριών που έχουν να κάνουν με τους δικαιούχου, τους πραγματικού. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το θέλει ούτε αυτό ο εισήγητη. Βεβαίω πρόκειται για σημαντικό σημείο το οποίο ε, εγκρίθηκε στην εκθεσμή του Ντάν για το εξέλιμα χρήματο. Οπότε η πράσινη θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει εδώ μια συνέπεια μεταξύ των δύο εκθέσεων. Γι' αυτό θα πρέπει και η ΕΤΕ να αναλάβει τι ευθύνε τη όσον αφορά αυτές τις προσπάθειες ε, καταπολέμησης του, του ξεβλήματος χρήματος. Αυτά γιατί δεν μπορούμε ε, στη μία περίπτωση να επιψηφίζουμε κάτι για να καταψηφίζουμε στην άλλη. Αυτό δεν είναι συνέπεια. Εν κατακλείδη να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πρέντα της μας των Πρασίνων για το έργο το οποίο επιτέλεσε Αυτά. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο εις τους άλλους συναδέλφους, εάν θέλετε το λόγο, για τις εγγύσεις της Ένωσης προς την ΕΤΕ. Τότε κύριε Πρόεδρε, να σας δώσω ξανά τα πράγματα. Ο κύριος Πρέντα. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτό το οποίο μου είπατε για τις συμβαστικέ ε, τροπολογίες στις οποίες κατέληξα. είναι πολύ σημαντικά. Ε, δεν μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε επί όλων. Πότε και πάμε στην ψηφοφορία και θα δούμε. Εγώ εμένω στην απόψή μου το άρθρο 42 ή 30, 43. εγώ το 33 προτείνω χωρίς την ψηφορία. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε να διευκρινίσουμε τη θέση κάθε πολιτική ομάδα. Πάντω θέλω πάντα να σα ευχαριστήσω για τη συνεργασία του Πρασίνου. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο, και σας υπενθυμίζω ότι η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα κιόλα. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε για τη γραμματεία μας. Και όλους όσους τοποθετήθηκαν. Τώρα, για να το σημείο παρελθόν 12 σημερινή διατάξεω. Πρόκειται για ανταλλαγή από. Πρόκειται για την ετησία έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. δούμε δικαιώματα στον κόσμο 2012 και σχετική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόκειται για έκθεση του κυρίου Γκούσταψον, ο οποίο και θα δώσει τον ευκαιρίο ελάχισμα στην συζήτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπόρεσα να έρθω. Ενωρίτερα είχα άλλη ανηλυμένη υποχρέωση εδώ εντός του Κοινοβουλίου που ήταν σημαντική για την, ε, και για την Επιτροπή μας. Η έκθεση είμαι βέβαιος ότι θα αποβεί πολύ καλή. Λίγες τροπολογίες κατατέθηκαν για την έκθεσή μου, τις οποίες επιθυμώ να εξηγήσω, για παράδειγμα για την υπηρεσία εξωτερικών ε, δράσεων και τις αρμοδιότητές της. Είπατε επίσης και εσείς ότι όλες οι πολιτικές μας και στρατηγικές πρέπει να βασίζονται στην σωστή τήρηση των διατάξεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όπου και να βρισκόμαστε πρέπει να φροντίζουμε να γίνεται αυτό. Και αυτά πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη. Να εξασφαλίζουμε ώστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, η ισότητα των φύλων και τα σχετικά θέματα να διέρχονται σαν ερυθρό νήμα όλες τις πολιτικές της Ένωσης. Εγώ λοιπόν τώρα έχω καταθέσει πέντε τροπολογίες, πέντε ε, θέματα και νομίζω ότι χρειαζόμαστε εργαλεία για να εξασφαλίσουμε αυτή την προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να εφαρμόζονται παντού. Είναι σημαντικό στην εργασία μας να περιλαμβάνουμε και να, να, να προβαίνουμε δηλαδή σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, διότι αυτοί θα μας δώσουν τις απαραίτητες προφορίες. Εξάλλου είναι αυτοί που έχουν τις ειδικές γνώσεις. Πρέπει να τους δώσουμε λοιπόν περισσότερη προσοχή. Εμείς βέβαια είμαστε αυτοί που λαμβάνουμε τις αποφάσεις. Όμως η κοινωνία των πολιτών μπορεί να συμβάλλει σημαντικά διότι τα πρόσωπα αυτά έχουν λεπτομερείς γνώσεις των θεμάτων, λεπτομερή μάλλον γνώση των θεμάτων που δεν είναι δυνατόν να έχουμε για όλα τα θέματα εμείς και σε όλα αυτά τα επίπεδα. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δώσει υψηλή προτεραιότητα σε διαφόρους τομείς με ειδικού στόχους. Για παράδειγμα, συνδυασμό περιβαλλοντικών θεμάτων και θεμάτων κλίματος με κοινωνικά. Και πέρα το 2015. Αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση και νομίζω ότι ε, καλά κάνουμε. Πρέπει να συνδυάζουμε τους τομείς πολιτικής, διότι αυτοί αλληλοεπηρεάζονται. Συχνά η οικονομική δραστηριότητα επηρεάζει το περιβάλλον και το περιβάλλον με τη σειρά του την κοινωνία, την κοινωνική ζωή, ιδιότερα, ιδιαίτερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Υπάρχει και ένα, μια παράγραφο στο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών. Έχω περιλάβει σχετικές διατάξεις παλαιότερα. Εδώ όχι. Πέντε τροπολογίες έχουν κατατεθεί στο βασικό κορμό της έκθεσης που δεν είναι δικές μου. Θα ήθελα ωστόσο να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων μου. Ε, ευχαριστώ 300 άνθρωποι χάθηκαν έξω από τη Λαμπεντούζα πριν από λίγες μέρες. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καυτό θέμα. Ο κ. Μαρτίνες θέλει να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα με τη σειρά μου να δηλώσω την συμφωνία μου με τον κύριο Γκούστασον. Συμφωνώ για την κρίση του, για το περιεχόμενο της ε, εκθέσεως που συζητούμε και συμφωνώ και με αυτό που είπε η Πρόεδρος. Η τραγωδία της Λαμπεντούσα πιστεύω ότι αξίζει τουλάχιστον να υψώσει τη φωνή της η Επιτροπή μας. Πρώτον, διότι η έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών προηγήθηκε των συμβάντων της Λαπεντούσα, αλλά είναι σαφώς, συνδέεται σαφώς με τα θέματα της ανάπτυξης. Επίσης θα ήθελα να γίνει ένα σχόλιο για το θέμα αυτό από εμά που βρίσκω ότι είμαστε αρμοδιότεροι των συναδέλφων της Επιτροπής Εξωτερικών. Είναι κάτι που μας απασχολεί Πρωτίστως, είμαι βέβαιος ότι ως εισηγητής ο κύριος Γκούσταυσον θα κάνει συστάσεις πρόσθετες έτσι ώστε η Επιτροπή Εξωτερικών να μπορέσει να περιλάβει στο κείμενό της μια έκκληση σαφή έκκληση διότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει καρφωθεί στη συνείδηση εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Για τη Λαμπεντούζα οι άνθρωποι στην Ιταλία και αλλού, σε όλη την Ευρώπη έχουν αγανακτήσει γιατί έχουν την εντύπωση ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν προχωρεί τίποτα. πέρα από τις προσευχές για τις ψυχές των απολεσθέντων, αλλά ως πολιτικοί έχουμε κάποια ευθύνη. Να υψώσουμε τη φωνή μας, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει για να μην συμβούν τέτοια πράγματα ξανά στο μέλλον. Ήδη η Ιταλική κυβέρνηση, νομίζω, έχει αποφασίσει να λάβει μέτρα. Αναμένω να δω τα μέτρα αυτά, αλλά χωρίς πολύ πεποίθηση. Τι θα κάνουν, θα κινητοποιήσουν ακόμα περισσότερο τα πολεμικά σκάφη για να απομακρύνουν αυτούς που προσπαθούν να προσεγγίσουν τις ακτές. Μα δεν πρόκειται γι' αυτό. Δεν πρέπει εκεί να κατευθύνουμε τις προσπάθειές μας. Έχω ωστόσο εμπιστοσύνη στον εισηγητή και θα τον παρακαλέσω ως εισηγητής, ο κ. Γκουσταύσον, να υποβάλει το συντομότερο δυνατό μία-δύο παραγράφους με τις οποίες να εκφράζουμε την αρισχία μας, την αλληλεγγύη μας και την ανάγκη να αναλυθεί δράση. Σεις κύριε Κόρτες Λάστρα. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Γκούσταυσον και να σας πω μια σύντομη σκέψη μου. Ακριβώς όπως είπε και ο Μιγελάχελ Μαρτίνεθ ότι όντως πρόσφατα δεν, έχω, δεν νομιμοποιούμεθα να μιλούμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα θα πρέπει να ζητήσουμε το πρόβλημα της Λαμπεντούζα. Να τώρα είπαμε για αυτό, αυτή την ελληνική συμφωνία πριν από λίγο, αλλά από την άλλη μεριά, την σημερινή μέρα, δεν έχουμε πλέον την νομοποίηση να λέμε το δικαιώματα, όπως είπατε και εσείς, για τη γνωστή υπόθεση Λαμπεντούζα. Είδατε επίσης πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε άνοδο των εξτρεμιστών που δεν σέβονται τα δικαιώματα. Είδατε τι γίνεται με τους Τσιγκάνου. Τι γίνεται σε διάφορες χώρες που σε όλους τα δικαιώματα, όπως είπε και ο κύριος Γκούσταυσον, ε, τα είπε καλά, αλλά να λάβετε υπόψη επίσης και τη δική μου σκέψη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να πω και εγώ κάτι. Θα ήθελα να ζητήσω τη Γραμματεία να εξετάσει το ενδεχόμενο διοργάνωση για την Επιτροπή Ανάπτυξης αντιπροσωπείας που να μεταβεί στη Λαμπεντούσα γρήγορα αν είναι ακόμα δυνατόν, αν δεν έχουμε πλέον χώρο ή χρήμα, στο το διοργανώσουμε με τους δικούς μας πόρους, ούτως ώστε η Επιτροπή Ανάπτυξης να είναι παρούσα στρατικό τόπο για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό είναι κάτι πρέπει να το συζητήσουμε με τους συντονιστές και να δούμε μήπως μπορούμε να θέσουμε και προφορική ερώτηση με ψήφισμα στην επόμενη σύνοδο της Ολομέλειας στο Στρασβούργο. Κύριε Γκούσταυσο, να παραμείνουμε σε επαφή για να προχωρήσουμε. Για την έκθεση για το σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είναι κάτι σημαντικό. Αλλά να δείξουμε και με την επικαιρότητα αυτή που είναι ένα φαινόμενο πραγματικά δυσβάσταχτο, απαράδεκτο. Να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκπρόσωπος για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης είναι η κυρία Τίσον που την εκπροσωπεί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την παρέμβασή του και για τα όσα προτείνει. Λέει ότι σημειώνουμε ότι θα πρέπει περί εξωτερική δράση να υπομειστεί περισσότερε ευθύνε όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα πλαίσια και το σεβασμό του όταν αναφέρεται στη συμπερίληψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλε τι πολιτικέ, αυτό είναι κάτι προβλέπεται στη στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία που θετήθηκε τον Ιούνιο του 2012 και στο σχέδιο δράση, που ακολούθησε. Τέταρτο κεφάλαιο τη στρατηγική που συμπεριλαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα εσωτερικά και εξωτερικά και το σχέδιο δράση, υπαριθμών 10 δράσει σχέδιο δράσης για να υπάρξει μια προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλε τι αναπτυξιακέ πολιτικέ και θα παραθέσω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Όταν προτείνεται τροπολογίε, λέτε ότι πρέπει να υπάρχει ένα σύνολο εργαλείων που θα επιτρέπει προσέγγιση βάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύνολο εργαλείων που αναπτύξαμε τον περασμένο χρόνο. Επίσης έχουμε αναπτύξει και ένα έγγραφο, μία έννοια, μία προσέγγιση, έγγραφο εργασίας, επεξεργαζόμαστε και ολοκληρώνεται από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΤΕΦΚΟ. Συνεργαζόμαστε με την ΤΕΦΚΟ. Θα υπάρξει συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Μερίδα Ανάπτυξη, θα υπάρξει ένα πάνελ ακριβώ με αυτό το θέμα, πώ τα ανθρώπινα δικαιώματα θα συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα ψηφιακά θέματα. Και στα πλαίσια του Φόρουμ των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Δεκεμβρίου και εκεί θα συνεργαστούμε και με την κοινωνία των πολιτών. Λοιπόν, όσον αφορά συγκεκριμένο επίπεδο, ήδη πέρσι υιοθετήσαμε στα πλαίσια της οικονομικής υποστήριξης υιοθετήσαμε μια προσέγγιση με προσανατολισμούς σχετικά με το πώς οι χώρες ακολουθούν και εφαρμόζουν τις θεμελιώδεις αρχές, εισέβονται τις θεμελιώδεις αρχές, υπάρχει μεθοδολογία για τη γενική δημοσιονομική υποστήριξη, η τομεακή αυτή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ πολύ. Ξαναδεί το λόγο στον κύριο Γκούσταυσον για να ολοκληρώσουμε το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και εγώ συμφωνώ με τις ανησυχίες που ξεφράστησαν. Συμφωνώ και με τα σχόλιά σας για τη Λαμπεντούσα και τα όσα είπε ο κύριος Κορτές και άλλοι και ο κύριος Μαρτίνες. Όπως είπε λοιπόν ο κύριος Κορτές, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να χάσουμε την αξιοπιστία μας και την νομιμότητά μας όσον αφορά τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων εάν θεωρεί ο κόσμος ότι έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δράσουμε. Και νομίζω ότι είναι κάτι που θα έπρεπε να το προσθέσουμε εδώ στη συγκεκριμένη γνωμοδότηση, κάτι που σχετίζεται με τη Λαμπεντούσα. Να πω επίσης και κάτι άλλο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τα διάφορα εργαλεία της εργαλειοθήκης. Υποθέτω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι καλό το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία της εργαλειοθήκης. Ενισχύεται έτσι η εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τους βοηθάμε σε αυτό που κάνουν. Να πω επίσης ότι συμφωνώ αληθεύει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πάντα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις αναπτυξιακές πολιτικές. Σε διάφορα έγγραφα πολιτικής αναφέρεται αυτό. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως. Δεν είναι το τι αναφέρεται στα έγγραφα. Το θέμα είναι πώς εφαρμόζονται. Αυτό ισχύει για πολλές πτυχές του έργου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όπως η ισότητα των φύλων. Κάτι με το οποίο ασχολούμαι αρκετά. Αναφέρεται στη συνθήκη της Λισαβόνας σε διάφορα έγγραφα πολιτικής δεν είναι εδώ το πρόβλημα. Πολύ συχνά το πρόβλημα είναι ότι δεν εφαρμόζεται η αρχή σωστά και δεν διατίθενται πόροι που επιτρέπουν την εφαρμογή της αρχής. Άρα δεν αρκεί να λέμε κάτι, να λέμε ότι είναι σημαντικό και να συμφωνούμε. Πρέπει να υλοποιούμε αυτά που λέμε. Οι δράσεις μιλούν περισσότερο από τα λόγια, έτσι μπορεί να δείξει κανείς ότι παίρνει κάποια πράγματα στα σοβαρά. Θα σας ευχαριστήσω όλους και ζητώ συγγνώμη που θα φύγω, αλλά προεδρεύω ε, μια άλλη συνεδριάσεω, οπότε πρέπει να αποχωρήσω. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Θα συνεχίσουμε λοιπόν το σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης που αφορά την μείωση των κινδύνων, καταστροφών Είχαμε τη συμμετοχή της, ε, της Επιτρόπου Γιώργεβα και της ειδική εκπροσώπου της υπεύθυνη από πλευρά Γενικής Γραμματείας του ΟΗΕ όσον αφορά την ανθεκτικότητα και τιμή των κινδύνων καταστροφών ε, για τη συζήτηση. Θα συζητήσουμε λοιπόν την έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής μας για το ίδιο θέμα, δηλαδή την ανθεκτικότητα και τη μείωση των κινδύνων καταστροφών. Ο κύριος Γκέι Μίτσελ είναι εισηγητής μας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συνάδελφοι, τον περασμένο Οκτώβριο εξεδήλωσε ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ενώσης όσον αφορά την ανθεκτικότητα μαθαίνοντας από την κρίση ασφαλείας των τροφίμων αυτή η ανακοίνωση θέλει να δώσει κατεύθυνση στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας και τη μείωση του ευαλότου χαρακτήρα των διαφόρων αναπτυσσομένων χωρών, κυρίως εκείνων που αντιμετωπίζουν περισσότερες κρίσεις. Εγώ εδράζομαι όχι μόνο επί της προσεγγής Ευρωπαϊκής Ενώσης για την ανθεκτικότητα, αλλά επί τη σημαντικότητα της συνιστώσεως της ανθεκτικότητας, δηλαδή μείωση του κινδύνου καταστροφών, με αρχικά αγγλικά DRR Λοιπόν, είχαμε ανακοίνωση επενθεκτικότητα και ακολούθησε το σχέδιο δράση για την ανθεκτικότητα των χωρών που αντιμετωπίζουν κρίσει 2013-2020. Η έκθεσή μου έλαβε υπόψη αυτό το σχέδιο δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τόνισε ότι οι προτάσει και οι προτεραιότητε που αναφέρονται θα πρέπει να εφαρμοστούν αποτελεσματικά και ότι συνεχής πρόοδο θα πρέπει να εφαρμόζεται για την επίτευξη των στόχων. Το Σεπτέμβριο 16 Σεπτεμβρίου φέτος, όπως είπατε κυρία Πρόεδρε, έγινε ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο για Ανθρωπιστική Βοήθεια, την Επίτροπο Γεώργεβα και εσεί και ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας για την μείωση του κινδύνου καταστροφών, ειδικό εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα, της, Γενικούς Γραμμα... της Γενικής Γραμματέας Μάργαρετ Galston όσον αφορά την ανθεκτικότητα και μείωση του κινδύνου μετά το 2015 και το σχετικό πρόγραμμα. Σημαντικότατη ήταν αυτή η εκδήλωση που μας βοήθησε να πλησιώσουμε πολλά ουσιαστικά πράγματα και ιδέες εκθέσεως. Η Επίτροπος κυρία Γεωργίευα πρότεινε ότι η έκθεση θα πρέπει να εστιάζεται επί των πλέον ευαλώτων ατόμων και κοινοτήτων και είχαμε σαν στόχο να κάνουμε ακριβώς αυτό για να βελτιωθεί η προσέγγιση για την ανθεκτικότητα, η καλή έκθεση για σημαντική ενσωμάτωση μέτρων ανθεκτικότητας στην αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια και προγραμματισμό. Η έκθεση αναγνωρίζει επίσης τις προκλήσεις που δημιουργούνται από την αλλαγή του κλίματος. Τονίζει επίσης ότι η αλλαγή του κλίματος και οι σχετικές προσαρμογές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην ανθεκτικότητα και τις διάφορες πρωτοβουλίες DRR για τη μέση του κινδύνου καταστροφών. Ο αντίκτυπος των καταστροφών ε, οδηγεί σε σημαντικές οικονομικές ε, απώλειες για πληθυσμούς και κυβερνήσεις καθώς και τεράστιες απώλειες ζωών, έτσι σημαντικότερο. Λοιπόν, πρέπει να αναλύσουμε και να διαχειριστούμε καταστροφές για να μειώσουμε τον, ε, το ευάλωτο στις καταστροφές οικοδομώντας ανθεκτικότητα. Καλύπτονται δραστηριότητες οι οποίες υποστηρίζουν την προετοιμασία, την πρόληψη και την μείωση των συνέπειων από τοπικό μέχρι διεθνές επίπεδο. Αυτή η έκθεση τόνισε το ότι η επένδυση σε μέτρα μείωσης των κινδύνων πριν τις καταστροφές είναι πολύ πιο αποτελεσματικό όσον αφορά το κόστος από τη χρηματοδότηση, ανταπόκριση σε καταστροφές μετά την εκδήλωση της καταστροφής. Η Ιατρική Τράπεζα Ανάπτυξη εκτιμά ότι ένα δολάριο που επενδύεται για τη μείωση του κινδύνου από καταστροφέ σε περιοχέ που αντιμετωπίζουν κρίσει εξοικονομεί τουλάχιστον 4 δολάρια όσον αφορά την αποστολή βοήθεια και τι προσπάθειε ανοικοδόμηση και το σχετικό κόστο στο μέλλον. Από ό,τι καταλαβαίνω, 3 δισεκατομμύρια που δόθηκαν στην Κίνα, ακριβώ αυτό πέτυχαν. Ε, γλιτώσαμε πάνω από 12 δι και ζωέ βέβαια και καταστροφέ που προλάβαμε. Λοιπόν, η έκθεση καθιστά σαφέ ότι η μείωση του κινδύνου καταστροφών πρέπει να έχει προτεραιότητα σε μελλοντικό προγραμματισμό για την ανάπτυξη και θα πρέπει να συνωματώνεται και σε αναπτυξιακή βοήθεια και ανθρωπιστική βοήθεια και σχετικό προγραμματισμό σε όλε αυτέ τι χώρε. Έτσι, δε περαιτέρω, ζητά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλου σχετικού φορεί να συμπεριλάβουν τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και τι προσαρμογέ και τι στρατηγικέ την του κλίματο και να συντονίζονται οι προσπάθειε για να αναρμονίζονται αυτέ οι δραστηριότητε. Η έκθεση αναγνωρίζει την καλή δουλειά που έκανε το πλαίσιο του ΟΕΕ για τη δράση στο δεκαετές πλαίσιο που εκμένει το 2015 και τόνισα ότι ε, το μετά το δημοσιονομικό πλαίσιο, το σχετικό πλαίσιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα του πλαισίου εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι μετά το 2015 το πρόγραμμα θα θα ενσωματώνει την μείωση του κινδύνου καταστροφών και την αθεκτικότητα. Η ανάπτυξη αθεκτικότητας και η πρόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης απαιτεί μια προσέγγιση κοινωνική, τοπική, τοπικές αρχές, αρχές εκπροσώπους των πολιτών, πολίτες, μη κυβερνητικέ οργανώσεις και αναπτυξιακού εταίρους. Ο στόχος της εκθέσεώς μας είναι να τονίσει τη σημασία που έχουν όλοι οι φορείς για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας, κυρίως οι τοπικοί φορείς που μπορούν να παίξουν κεντρικό ρόλο και να συντονίσουν και να υποστηρίξουν πολυεπίπεδη προσέγγιση πολλαπλών φορέων για να απτυχθεί ανθεκτικότητα και η αρχή τη πρόληψη του κινδύνου καταστροφών. Είναι σημαντική αυτή η προσέγγιση ανθεκτικότητα να οδηγεί σε βιώσιμα ωφέλη για τι πλέον ευάλωτε περι... ε, κοινότητε τη κοινωνία, κυρίω εκείνου που ζουν σε ακραία φτώχεια και σε φτωχογειτονιέ, σε προχειρόσπιτα κλπ. Και που αντιμετωπίζουν πολύ ε, μεγάλο κίνδυνο. Οι αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως αυτές με πολύ χαμηλό εισόδημα, εκεί πολλά νοικοκυριά ζουν συνεχώς σε μια κατάσταση φτώχειας. Και εκεί έχουν ελάχιστη και μηδαμινή ε, κοινωνική προστασία. Άρα εκτίθενται πολύ περισσότερο στις καταστροφές. Γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε την κοινωνική προστασία που παρέχουμε σε αυτούς και τις διάφορες πολιτικές ασφάλισης αναπτυσσόμενες χώρες, ένα θέμα που έχουμε συζητήσει σε άλλο πλαίσιο. Είναι σημαντικό επίση, Πρόεδρε, αυτή η έκθεση να ασχοληθεί με την επιστημική ασφάλεια στα πλαίσια τη ανθεκτικότητα και τη πρόληψη του κινδύνου καταστροφών, κάτι που ήδη τόνισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι καταστροφέ και οι κατεπίγουσε ανάγκε πολύ συχνά ακολουθούνται από επιστημική κρίση και κακή διατροφή των διαφόρων πληγέντων πληθυσμών αυτή, όταν συμβαίνουν αυτές οι κρίσεις επιστημιστικές που δημιουργούνται από φυσικές ε, ή ανθρωπογενείς καταστροφές, αυτό είναι ένα φαινόμενο που όλο και αυξάνεται από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Είχαμε 50 με 65 επιστημιστικές ανάγκες το χρόνο από το 2000. 25 με 45 έγιναν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90. Οι φυσικές καταστροφές καταστρέφουν τη γεωργία και τις θετικές υποδομές ε, και τα στοιχεία ενεργητικού, τις οδιές, την παραγωγή, τη δυνατότητα παραγωγής. Αυτή η έκθεση τονίζει ότι η προσέγγιση ανθεκτικότητα πρέπει να εστιάζεται επί τη αύξηση επιστημιστική ασφάλεια και τη διατροφή και θα πρέπει συστηματικά αυτέ οι αρχέ να σηματώνονται στι διάφορε αποφάσει περί προγραμματισμού. Αρκετέ μελέτε έχουν εκπονηθεί και έχουν καταδείξει ότι σημαντικές οικονομίες μπορούν να επιτευχθούν αν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη μπορούν να συντονίσουν την αναπτυξιακή τους πολιτική και την ανθρωπιστική τους πολιτική και δραστηριότητα καλύτερα. Οι προσπάθειες για ανθεκτικότητα θα πρέπει να συντονίζονται πάρα πολύ μεταξύ κρατών μελών διεθνών οργανώσεων, δημοσίων θεσμών και κυρίως μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα πρέπει να συνεργάζονται και ο ιδιωτικό τομέα, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, η κοινωνία των πολιτών μπορούν όλοι αυτοί να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Αυτή η έκθεση θεωρεί και φρονεί ότι θα πρέπει να καταβληθούν σημαντικέ προσπάθειε για να αντιμετωπιστούν οι ανεπαρκή χρήση τη χρηματοδότηση για τη μείωση κινδύνου καταστροφών και τη ανθεκτικότητα και επικάλυψη προσπαθειών των σχετικών. Εν κατακλείδη, κύριε Πρόεδρε, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διεθνεί οργανώσει μπορούν να σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά τη μίση του κινδύνου καταστροφών και την ανθεκτικότητα στι αντισόμενε χώρε και στα προγράμματα που εφαρμόζουν εκεί. Είναι πρωταρχική όμω ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των πολιτών του. Γι' αυτό οι χώρε εταίροι θα πρέπει να έχουν πολιτική δέσμευση, την υποστήριξη και εφαρμογή δραστηριοτήτων οι οποίε διευρύνουν την ανθεκτικότητα και τη μείωση κινδύνου καταστροφών. Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση είναι σημαντικότατη και είναι μια δυνατότητα η θέση του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτού τη ανακοινώση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ενώση Ανθεκτικότητα να επιτευχθεί. Αυτή καθ' αυτή η προσέγγιση είναι τεράστιο κομμάτι τη αναπτυξιακή πολιτική. Ελπίζω ότι αυτή η έκθεση θα μπορεί να ενθαρρύνει αυξημένη υποστήριξη για την ανθεκτικότητα και τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και των συναφών δραστηριοτήτων και ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να προωθούμε αυτά τα θέματα, κυρίω όσο προσεγγίζουμε την περίοδο που ακολουθεί το 2015. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πολύ αγαπητοί κύριε. Η κυρία Χολ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη από τον εισηγητή γιατί σε λίγα λεπτά πρέπει να αποχωρήσω, να πάω σε άλλη επιτροπή. Βρίσκω όμως την έκθεσή του θαυμάσια. Έχει ευρύ φάσμα, καλύπτει πολλά σημαντικά θέματα, την σημασία συντονισμού ανθρωπιστικής πλευράς με την πλευρά της ανάπτυξης. Ίσως σε ορισμένα μπορούμε να προχωρήσουμε κάπως περισσότερο. Ο κύριος Μίτσελ τόνισε τον ρόλο των ε, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Εδώ ίσως πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση. Ιδίως σε εύθραυστες χώρες όπου δεν υπάρχει επαρκής ε, υποδομή, ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών μπορεί να αποβεί σημαντικός για την επιβίωση των κοινωνιών μετά από θεομηνίες, καταστροφές και για να αναπτύξουν μια ανθεκτικότητα. Είπε επίση ο κύριος Μίτσελ πόσο σημαντική είναι η διασύνδεση μεταξύ θεομηνιών και της εξασφάλισης των προστοζήν. Είναι η μεγάλη σημασία των μικρών καλλιεργητών, είναι μεγάλη και η σημασία των μικρών κτηνοτρόφων Υπάρχει και σχετική έκθεση για τους μικρούς βοσκούς κλπ. Και η έκθεση αυτή με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο μπορούν αυτοί οι μικροί κτηνοτρόφοι να εξασφαλίσουν τα ίδια τροφής που είναι απαραίτητα για, του, για τις τοπικές κοινωνίες, όχι μόνο με την παραγωγή κρέατος αλλά και γάλακτος αίματος και άλλων σχετικών. Είναι σημαντικό αυτό για την επιβίωση των τοπικών κοινωνιών. Τέλος, ναι μεν η έκθεση αυτή αναφέρεται ιδίω στην προοπτική των αναπτυσσόμενων χωρών και την αντιμετώπιση εκεί των θεομηνιών, αλλά ας μην δυσμονούμε όμως τον ρόλο που μπορούν να παίξουν και οι ανεπτυγμένες χώρες. Πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια μείωσης των αρνητικών συνεπειών της αλλαγής του κλίματος και ό,τι κάνουμε εμείς από τη δική μας πλευρά ως χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέεται σημαντικά με την ικανότητά μας να μειώσουμε την, τον κίνδυνο που προκύπτει από ενδεχόμενες θεομηνίες σε αναπτυσσόμενες χώρες. Υπάρχει λοιπόν ένα σύνδεσμος μεταξύ αυτών των δύο παραγόντων που αποδεικνύεται όλο και περισσότερο αν είδατε και την έκθεση της ICC προ λίγων ημερών. Ευθύνη φέρουμε επίσης για την χρηματοδότηση, διότι είπαμε ότι θα δίνουμε μέχρι το 2020 100 δισεκατομμύρια τον χρόνο και πρέπει όντως να τα δώσουμε τα λεφτά αυτά. Βρίσκω ότι είναι, είναι σημαντική και ε, εξαιρετική η έκθεση αυτή και θα μας απασχολήσει και άλλο. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ντέβα. εγώ δεν επρόκειτο να πω «Α, υπάρχει κάποια σύγχυση». Όχι εσάς. Ο κύριος Δέβα ε, προηγείται. Τότε να μην πω τίποτα. Καλά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, λέει ο κύριος Ντέβα. Ας αρχίσω συγχαίροντας τον κύριο Μίτσελ για την θαυμάσια έκθεσή του. Έχω την ατυχή εμπειρία να ειδώ το τσουνάμι στη Σρι πάνω από ένα μπαλκόνι. Προκαιρού κατάφερα να αναλύσω τι ακριβώς γίνεται αν ταξινομήσει κανείς τις θεομηνίες σεισμοί, τσουνάμι, παλιροϊκά κύματα, δηλαδή κατολιστήσεις πλημμύρες, κατολιστήσεις, ε, κατολιστήσεις λάσπης. Αυτά είναι, αυτές είναι οι πιο μεγάλες ε, καταστροφές που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις καταραίουν τα κτίρια και μετά την κατάρρευση των κτιρίων Πρωταρχικό ρόλο έχει μετά η αποκομιδή αυτών των ε, ερηπείων. Χρειάστηκαν εκεί μετά από το παλιροϊκό κύμα 18 μήνες μέχρι ότου καθαριστούν όλα αυτά τα ερήπια. Από τα άμεσα πράγματα λοιπόν που πρέπει να προσφέρει ανακουφιστική βοήθεια τρόφιμα, νερό, είναι να ανοίξουν οι δρόμοι για να φτάσουν αυτά τα πράγματα στους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Το ίδιο έγινε στο Παγκλαντές, χρειάστηκαν 8 μέρες για να σκάψουν υπό τα ερήπια και βρήκαν και μάλιστα ένα νεαρό άτομο που είχε επιβιώσει 8 μέρες μετά. Γιατί χρειάστηκαν τόσο χρόνο, θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς, για να σηκώσουν μερικά κομμάτια μπετών. Η απάντηση είναι απλή οι χώρες αυτές δεν έχουν τα βαριά μηχανήματα γερανούς και άλλα που μπορούν ε, να το κάνουν. Ο καλύτερος τρόπος για να πάνε τα μηχανήματα αυτά εκεί είναι ελικόπτερα μεγάλων φορτίων. Ο το ίδιο για τις πλημμύρες του Πακιστάν, όπου ε, πλήγησαν 14 εκατομμύρια άνθρωποι. κατέρευσαν οι αιστείες τους, έχασαν τις αιστείες τους, κατέρευσαν τα, τα σπίτια τους. Οι Πακιστανοί είχαν τη δυνατότητα, είχαν τα μηχανήματα για να κάνουν αυτή την αποκομιδή, τέλο πάντων, να σηκώσουν αυτά τα κομμάτια τείχων κτλ. Άρα ένα σημαντικό στοιχείο είναι η ικανότητα να μπορούν να σηκώσουν ε, βαριά αντικείμενα και κυρίως με ελικόπτερα. Τώρα πώς θα φτάσουν τα ελικόπτερα εκεί μέσα σε 24 ώρες αυτό είναι άλλο θέμα. Ίσως στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση θεομηνιών πρέπει να σκεφτούμε πώς θα κατανείμουμε ελικόπτερα ανά τον κόσμο βέβαια και με ανθρώπους που να είναι ικανοί να τα χειριστούν. Είναι ένα ε, ε, βασικό πρόβλημα εφοδιασμού το οποίο θα ήθελα να απασχολήσει τον εισηγητή. Ο κ. Μέσερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα όσα είπαν οι προηγούμενοι. Είναι επιτυχής η έκθεση που έχει συντάξει ο κύριος Μίτσελ. Τώρα, οι στόχοι είναι δύο. Πρώτα, η ανθεκτικότητα των αναπτυσσόμενων χωρών για να αντιμετωπίζουν τέτοιες αμυνίες πρέπει να βελτιωθεί. Δεύτερο, οι αναπτυσσόμενες χώρες χρειάζονται την ενίσχυσή μας για να μπορούν να συνέρχονται μετά από κρίσεις τροφίμων. Εκτός από την ταχεία βοήθεια που πρέπει να δοθεί, είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι αιτίες να αναλυθούν και να ληφθούν διαρθρωμένα μέτρα. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Αφενός υπάρχει η πρωτοβουλία SHARE που προβλέπεται για το κέρας της Αφρικής και επίσης για τη ζώνη Σαχέλ η πρωτοβουλία Άτζια. Το SHARE για το κέρας της Αφρικής περιλαμβάνει για παράδειγμα σε βάθος ανάλυση των αιτίων, αξιολόγηση των παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθορισμό προτεραιοτήτων. Οι αιτίε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κέρας της Αφρικής, ως γνωρίζουμε όλοι, είναι η ασθενής πολιτική ηγεσία, η καταστροφή του περιβάλλοντος, συγκρούσεις για τους βασικούς πόρους όπως βοσκοτόπια και νερό και συγκρούσεις για τη χρήση της γης. Το άλλο υποδειγματικό εγχείρημα, άγια για την ζώνη Σαχέλ, βασίζεται σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης καθώς και παρακολούθηση των αγορών. Οι συγκομιδές της ζώνης Σαχέλ το 2013 ήταν καλές. Όμως τα προϊόντα ακρίβηναν για τα πιο ε, φτωχά νοικοκυριά. Μία από τις αιτίε των ξηρασιών είναι η αλλαγή του κλίματος. Εδώ χρειάζεται υπεύθυνη πολιτική πρόληψης καθώς επίσης και κονδύλια από το Global Climate Change Alliance. Πρέπει ωστόσο να ληφθεί φροντίδα οι στόχοι να τηρούνται και όταν παρεμβαίνουν ιδιώτες επενδυτές. Συγκρούσεις τώρα για τη χρήση γης και το νερό δεν επιτρέπεται να οξύνονται εφόσον παρεμβαίνουν και επιχειρήσεις. Πρέπει να βελτιωθεί η κοινωνική κατάσταση και να χρησιμοποιούνται οι περιβαλλοντικοί πόροι με τρόπο αηφόρο. Η έκθεση της Κομισιόν του περσινού χρόνου βασίζεται σε κοινοπραξία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων όπως η New Alliance for Food Security που άρχισε να λειτουργεί ήδη από πέρσι υπό την αιγύδα των ΗΠΑ. Όμως ασκείται και πολύ κριτική στο κόνσεπτ αυτό γιατί πολλοί από τους επενδυτές είναι πολυεθνικοί όμιλοι με την έδρα τους στις Πολιτείες όπως η Μονσάντο με τις, ε, με τις δραστηριότητες αυτών των ομίλων στην Αφρική πολλοί μικροί γεωργοί χάνουν τις εκμεταλλεύσεις τους ή τις δυνατότητες δραστηριότητας ή υπερχρώνονται. Το ίδιο ισχύει για την αγορά σπόρων το, που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν άπαξ μόνο. Οι μικροί γεωργοί που αναγκάζονται να ε, λειτουργούν δίπλα στις μεγάλες ε, εκμεταλλεύσεις δεν έχουν πια αρκετό νερό για να ε, ποτίσουν τις καλλιεργίες τους. Οι ιδιώτες επενδυτές βεβαίως είναι σημαντικοί και καλοδεχόμενοι. Δεν μπορούμε να αναμένουμε όμως η αγορά, οι αγορές δηλαδή, να αντιμετωπίσουν ορθά και να μοιράζονται τους δικούς μας και περιβαλλοντικού στόχους. Η κοινοπραξία δημοσίων και ιδιωτικών φορέων βέβαια μας επιτρέπει να επιβάλλουμε εμείς ορισμένες συγκεκριμένες απαιτήσει. Για παράδειγμα, να ζητηθεί από τις επιχειρήσεις να δημοσιεύουν τα επενδυτικά του σχέδια σε ειδικές πλατφόρμες ώστε να εξασφαλίζει τη διαφάνεια. Από την προηγούμενη ισομερή συνέλευση ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης είδα ότι πολλοί Αφρικανοί παραπονέθηκαν ότι συχνά τους λείπει η πύρα και οι πόροι για να εξετάσουν τις συμφωνίες με Ευρωπαίους φορείς, ευρωπαϊκούς φορείς. Στόχος όμως της προαναφερθής συμμαχίας είναι και αυτός. Να δώσω ένα μικρό επιχείρημα, ένα μικρό παράδειγμα. Πρόκειται για την Ιάν Γκαμάρη από την Κένια, κτηνοτρόφο, η οποία μίλησε με γνωστή δημοσιογράφο σχετικά με το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να ενωθεί η επίγουσα επιστημική βοήθεια με την αναπτυξιακή βοήθεια. Από όπου και να έρχονται τα χρήματα, μας είπε η κυρία Μάρη. Είτε προέρχεται από Ταμείο Αντιμετώπισης Θεομηνιών, είτε προέρχεται από Ταμεία Προσαρμογής στις Κλιματικές Αλλαγές, είτε από τον προπολογισμό για τη μείωση της φτώχειας. Σημαντικό για μας είναι να μπορούμε να ζήσουμε ανθρώπινα με ασφάλεια και αξιοπρεπώς. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τέιλορ. Α, σας ευχαριστώ. Ε, ζητώ συγγνώμη για ε, την διασύνη με την οποία πήρα το μικρόφωνο πριν. Δεν θα πω πολλά. Καλή έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Μίτσελ. για την ατζέντα μετά το 2015, την ατζέντα δηλαδή της ανάπτυξης, αρχίζει να διαφαίνεται μια συνένεση για την διασύνδεση των στόχων της αηφόρου αναπτύξεως με, την, ε, με το ξερίζωμα της φτώχειας. Νομίζω ότι η ιδέα αυτή της ανθεκτικότητας και της μείωσης των επιπτώσεων των θεομηνιών πρέπει να περιληφθεί μέσα στη διαδικασία αυτή, διότι μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για να επιτευχθούν υποθούμενοι στόχοι. Σας ευχαριστώ και πάλι λοιπόν για την έκθεσή σας. Θα την υποστηρίξω όταν ε, θα έρθει η ώρα. Ευχαριστώ αγαπητέ Γκέι. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οποία εκπροσωπεί η κυρία Ιονέτ ή ο κύριος η κυρία Ντομινίκ Αλμπέρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να μου επιτρέψετε όπως τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής σας να εκφράσω την εκτίμησή μου και εγώ για την έκθεση η οποία δίνει τη σωστή έμφαση στην ανθεκτικότητα βασιζόμενη στη λογική που χρησιμοποίησε και η Επιτροπή για το μεγάλο αυτό εργοτάξιο με μια ανακοίνωση που βασίστηκε στα διδάγματα από την κρίση, την επιστηστική κρίση που προωθεί την ευρύτερη αυτή ιδέα της ανθεκτικότητας και που φτάσαμε έτσι τώρα στην έκθεση της Disaster Risk Reduction. Επιτρέψτε μου να σας πω και ίσως εδώ υπάρχει και κάποιο συμβολισμός ότι η πρώτη ανάληψη υποχρεώσεως μετά από την σχετική, από το σχετικό έγγραφο του Ιουνίου με το Action Plan ήταν για τη μείωση των κινδύνων στο project του ειρηνικού. Σας δείχνει αυτό τι σημασία αποδίδουμε. Η μείωση λοιπόν αυτή των κινδύνων και για τον κίνδυνο προκύπτων από τι κλιματικέ αλλαγέ παίζει σημαντικό ρόλο και στο σχέδιο που εγκρίθηκε στα μέσα Ιουνίου μετά από την έγκριση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Να σημειώσω κάπως περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα σημαντικά θέματα που ε, ακούστηκαν στη συζήτηση. Πρώτα, όσον αφορά το τι θα γίνει μετά το 2015. Πράγματι, η Κομισιόν υποστηρίζει την συζήτηση μάλλον τρεις κοινέ συζητήσεις τριών ομάδων εργασίας του Συμβουλίου. Βίπι, CODEV και Κονόν. Η ανακοίνωση για μετά το 2015 είναι καθαρή. Η Κομισιόν ε, επιθυμεί να επιτύχει συνένεση ώστε να περιληφθούν οι στόχοι της χιλιετίας με αυτούς της ε, ανάπτυξης. Αυτά τα περιλαμβάνουν και τα συμπεράσματα του Συμβολίου. εν ώψη και του έθραυστου χαρακτήρα που απειλεί την ανάπτυξη πάνω από 50 χωρών. Ευχαριστώ επίσης που λάβατε υπόψη τον, την ανάγκη συντονισμού των χωρών μελών. Και αυτό περιλαμβάνεται στο Resilience Action Plan που έχει ως στόχο να συνδυαστούν οι προσπάθειες επιτόπου Επίσης τονίζεται και στις νέες διατάξεις για τον κοινό προγραμματισμό. Με στόχο 50 και παραπάνω χώρες, οι περισσότερες από αυτές χώρες που αντιμετωπίζουν κινδύνους από διάφορες θεομηνίες και τώρα βεβαίως βρίσκονται στο επίκεντρο της συζητήσεως. Κάτι το οποίο ήδη τονίστηκε στη συζήτηση, αλλά το τονίζω και εγώ με τη σειρά μου, είναι ο ρόλος των εθνικών κυβερνήσεων και των πολιτικών δεσμευσιών τους και ταυτόχρονα η υποστήριξη που μπορούμε να δώσουμε μέσω των προγραμμάτων μας στις κυβερνήσεις αυτές σύμφωνα με τις αρχές για την εμπλοκή μας σε εύθραστα κράτη ιδίως ξεκινώντας με τις πρώτες αυτές επαφές και να μην ε, ε, επέλθει οποιοδήποτε κίνδυνος από τις δραστηριότητές μας λαμβάνοντας υπόψη τον έφραυστο χαρακτήρα και τον κίνδυνο που ενδέχεται να προκαλέσουν θεομηνίες. Διότι οι θεομηνίες μπορούν να επιδεινώσουν σοβαρά τον ήδη έφραυστο χαρακτήρα ορισμένων κρατών. Παράδειγμα, IT. Για αυτό το λόγο πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο έθραυστος χαρακτήρας και η ανθεκτικότητα ως δύο διαστάσεις του ίδιου πράγματος και να ληφθούν υπόψη και οι, άλλες, και οι άλλοι παράγοντες, όχι μόνο οι συγκρούσεις αλλά και οι κτλ. Επίσης να σας υπενθυμίσω όσον αφορά τις ε, περιφερειακές προσεγγίσεις, share και agir, ότι είναι τμήματα της συνολικής προσέγγισης την οποία στείλουμε στα πόδια της εδώ, είναι περιφερειακές στρατηγικές οι οποίες εξετάζουν την ανάπτυξη, την ασφάλεια, λαμβάνουν υπόψη την τεράστια ανθρωπιστική προσπάθεια που γίνεται ε, στα μέρη αυτά του κόσμου. Όσον αφορά την κοινοπραξία δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, όντως αυτό είναι σημαντική πτυχή του έργου μας. Είμαι βεβαίω ότι γνωρίζετε ότι η Επιτροπή συντάσσει ανακοίνωση τώρα για την συνεργασία του ιδιωτικού τομέα. Και βέβαια οι παρεμβάσεις στις χώρες αυτές λαμβάνουν υπόψη και τις ανάγκες αυτές. Τούτων λεχθέντων Επιθυμώ να σας τονίσω και πάλι ότι η εργασία στον τομέα αυτό, στον τομέα αυτό έχει την έννοια να αποδώσουν τα πράγματα αυτά στην πράξη. Να περιληφθούν λοιπόν αυτές οι πτυχές της ανθεκτικότητας και στα, στον προγραμματισμό μας. Βρισκόμαστε τώρα στην κρίσιμη στιγμή της φάσης του προγραμματισμού για να αποδώσουμε τα υπεσχημένα και στις χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω πάλι το λόγο στον κύριο Μίτσελ για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να ολοκληρώσω πάρα πολύ σύντομα για να ευχαριστήσω πρώτα πρώτα τους συναδέλφους για τα ευγενή του σχόλια. Για μου πρόκειται κάτι ε, επί το οποίο εάν συνεργαστούμε θα πετύχουμε πολλά. Και από ό,τι βλέπω όλες οι πολιτικές ομάδες έχουν την βούληση να προχωρήσουμε. Η Φιώνα ανέφερε το ζήτημα των αναπτύσσεων χωρών και την ευθύνη που υπάρχει. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, διότι θα το λάβουμε υπόψη. Για αυτά τα οποία είπε ο κύριος ε, Ντέβα για τα ελικόπτερα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι κάτι που δεν το είχα υπόψη μου. Ε, μας είπε και για τη χρήση της γης, μας είπε και για τι εταιρικέ σχέσει με το δυτικό τομέα. Και ο κ. Τελεόρ επίση είχε δίκιο όταν μα είπε ε, για την εκρίζωση κατά πολέμηση τη φτώχεια. Πάρα πολύ βασικό αυτό. Ε, να, μην δούμε κατασταλτικά ούτω ή πίνου. Είμαστε πιο. Πρέπει πιο πολλέ πρωτοβουλίε. Η σημασία όλων αυτών, σύμφωνα με την Επιτροπή, είναι ότι ίσω πιο γρήγορα πλησιάζουμε προς το τι θα κάνουμε μετά το 2015. Και δεν μιλώ μόνο για το τι θα κάνουμε εμείς τα τρία θεσμικά όργανα, αλλά τι θα κάνουμε όλα τα θεσμικά όργανα σε σχέση με τον ΟΗΕ. Γιατί θα έχουμε τον Επίτροπο, θα έχουμε το Γενικό Γραμματέα εδώ, να τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Οι παρατηρήσεις σα ήταν ε, μεγαλόψυχες. Άρα α προχωρήσουμε με συνένεση. Ας ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια. Γιατί νομίζω ότι να κάνουμε αυτό πρέπει, αυτό θα αποδώσει. Κύριε Μίτσελ, σας ευχαριστούμε για την τόσο εξαιρετική σα έκθεση. Και τώρα, σας μενθυμίζω ότι η προθεσμία για την κατάσταση των τροπολογιών ε, είναι 15 δεκάτου στις 5 η ώρα. Αύριο δηλαδή και 5 δεκάτου θα γίνει η ψηφοφορία. Και τώρα. Θα πάμε στις ψηφοφορίες. Παρακαλώ, βγάλετε τις κάρτες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Να κάνουμε πρώτα πρώτα μία δοκιμή. Ψηφίζουμε. Monsieur Taylor, il n'a pas la carte. Uh, Κύριε κύριο Στέιλο, δεν την έχω μαζί μου, πρόεδρε, συμπαθάτε με. Καλά. Εσείς θα ψηφίζετε παραδοσιακά με το χέρι και θα μετράτε ψήφο σας. Έχουμε εννέα, όχι, έχουμε εννέα που δεν έχουν κάρτα. Να κάνουμε μια ψηφοφορία. Κακό. Οκ. Ok. Le vote est clos. Le vote est clos. C'est bon. C'est bon. Alors, nous allons voter euh, l'opinion de... Και τώρα θα ψηφίσουμε την έκθεση του κυρίου Ντέβα. Τροπολογία υπαριθμών 8. Χωριστή ψηφορία, το πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος. Τροπολογία 8, δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Με μία ψηφοδιαφορά. Πρώτη τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Εγκρίνεται. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά αποχές, κρίνεται, τροπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, τροπολογία 10, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. ψηφοφορίας. Αν δεν λειτουργεί το μηχάνημα, η συσκευή για την ψηφοφορία. Κύριε Βάγγελο. Μπορείτε να μας πείτε τι ψηφίσατε. Όχι ψήφισα. Λεκτός μικροφώνου. Άρα απορρίπτεται η διάταξη αυτή. Τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6. Υπέρ κατά αποχές. 7. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 13. Έλεγχος. Ψηφίζουμε για το 7. Εγκρίνεται τότε. Ψήφισε υπέρ ο κύριος Τέιλορ και εσείς κατά. 10 συν 1, 11 εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές δεν θα γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουν Πέρας. Δέκα 16. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονική επαλήθευση ηλεκτρονική για το 17 ψηφίζουμε C'est rejeté avec euh, égalité de voix. Amendement 10. 18. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21. Χωρίς την ψηφορία, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 22. Υπέρ, κατά, η Επαλήθευση. 22. Δημιουργική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Κάποιος δεν ψήφισε. Πέρας. Απορρίπτεται 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψήφισμα τώρα με ένα στο σύνολο του κειμένου υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική παλήθευση. Ψηφίζουμε. Πέρας. Μα συγκρίνεται με 21-3. Καμία εποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Τώρα θα εξαγάμε την ψηφοφορία όσον αφορά την γνωμοδότηση του κυρίου Πρέντα. Τροπολογία υπαρθμών ένα, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 28 εκεί ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική υπερθυμόν 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Υπερθυμόν 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπερθυμών 3 υπέρ κατά. Άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 33 χωριστή ψηφορία. Πρώτο τμήμα. Α, όχι. Α, όχι, όχι. Παρέλειψα το υπερθυμών 3. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33. Χωριστή ψηφορία, πρώτο τμήμα υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. 33. Δεύτερο τμήμα. Συγγνώμη γιατί το 32 κατέπεσε. Άρα τι θέλει να αρχίσουμε από την αρχή. 33 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Υπέρ. Κατά. αποχέ Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το είναι καταπίπτη. Και το 35 συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. Το βλέπω 37 υπέρ. Κατά. άποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ. Κατά. εποχέ, Απορρίπτεται. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. εποχέ, εγκρίνεται. 12 ε, υπέρ. Κατά. Αποχέ Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά αποχή και θα παλιδεύσουμε για το 42 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. και το πολύ, υπάρχει μόνο δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. 18. Και contre, qui s'abstient, Και το 18 εγκρίνεται και το 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική 3 υπέρ contre, qui s'abstient, adapté. Εγκρίνεται και υπαριθμών 20 και 4. Υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική υπαριθμών 5 υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική 6 εγκρίνεται. 25, 26 μάλλον, κατά 25, 26 εγκρίνεται και 27 υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται. Τροπολογία. προθεμόν 43 υπέρ Κατά. Α, όχι, όχι. Πρόκειται για το πρώτο τμήμα, πρέπει να το έχω διευκρινίσει, οπότε πάμε πίσω, ξαναρχίζουμε. Πρώτο τμήμα του 43, υπέρ. Κατά. Αποχίες. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα καταπίπτει. 44, υπέρ. Κατά. Αποχίες. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολία 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε τώρα το σύνολο τη γνωμοδοτήσεως όπως ε, έχει τροποποιηθεί με ένα χειρός υπέρ. Κατά αποχέ. εγκρίνεται. Και ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Ομοφόνος. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. aborde le point à l'ordre du jour. Πάμε στο 16. Πρόκειται για το πλαίσιο τη πολιτική που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια. Με ορίζοντα χρονικό το έτο 2030. Είναι το τελευταίο σημείο. Ε, το ουσιαστικό που έχουμε στη διάταξη. Θα συζητήσουμε γι' αυτό το σχέδιο νομοθετήσεως που αφορά ένα τέτοιο σχέδιο για τι πολιτικέ για κλίμα και ενέργεια με ορίζοντα το 2030. Ένβη και Ήτρα είναι οι συναρμόδιες επιτροπές. Η συγητής μας είναι ο κύριος Νόιζερ, εις τον οποίο και δίνω το λόγο μας παρουσιάσει το κείμενο του. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μετά από μια ψηφοφορία βέβαια, όπως στην Εκκλησία, μόλις ψάλουν τον τελευταίο ύμνο, πολλοί σηκώνονται και πάνε σπίτι τους. Όμως η έκθεση είναι σημαντική και η γνωμοδότησή μας δυστυχώς πρέπει να είναι, οφείλει να είναι πολύ σύντομη διότι πιο ε, αρμόδιες επιτροπές και πιο σημαντικές είναι ΕΝΒΙ και ήτρε. Παρ' όλα αυτά ίσως είναι πιο απλό να συντάξουμε τη γνωμοδότηση αυτή. Οι αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος πλήττουν κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες που είναι και εκείνες οι οποίες ευθύνονται λιγότερο. Ωστόσο υφίστανται κατεξοχήν τις βαριές συνέπειες. Εμείς ως βιομηχανικές χώρες έχουμε τη μεγαλύτερη ευθύνη και γι' αυτό είμαστε και εκείνοι που πρέπει να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο μειώνοντας τις εκπομπές μας. Προτείνω τρεις δεσμευτικούς στόχους για το 2030 μείωση των ε, εκπομπών αερίων κατά 50%, αύξηση των ανανεώσιμων ενεργειών κατά 40% και αύξηση της αποδοτικότητας χρήσης της ενέργειας στο 30%. Εκτός αυτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη θα πρέπει να καταργήσουν σταδιακά τις επιδοτήσεις για την εξόριξη ορυκτών φορέων ενέργειας. Νομίζω ότι χρειάζεται αλλαγή παραδείγματος εν προκειμένου. Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς της ενέργειας και η διαμεθοριακή διακίνηση της ενέργειας θα πρέπει να διευκολύνουν την ανταλλαγή ενέργειας. Επίσης, τα βιολογικά καύσιμα προκαλούν όλο και περισσότερα προβλήματα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Μετά το 2020 πιστεύω ότι δεν πρέπει να θεσπιστούν άλλοι στόχοι, άλλοι ευρωπαϊκοί στόχοι για τα βιοκαύσιμα. Ας υπενθυμίσουμε επίσης τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει χώρες μέλη για τις χρηματοδοτήσεις για την αντιμετώπιση των ε, αλλαγών του, κλίμακος, κλίματος και να μην συμψηφίζονται με τα χρήματα που δίνουν για ανάπτυξη. Βεβαίως είναι σημαντικό να υπάρχει πλαίσιο, λέει η Πρόεδρος, για τις πολιτικές του κλίματος και της ενέργειας με ορίζοντα το 2030. Ουδής επιθυμεί να λάβει το λόγο. Καλώς, συγχαίρω τον κύριο Νόισερ για την σημαντική έκθεσή του και δίνω το λόγο στην Κομισιόν. Ο κύριος Φεργουτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ ιδίως τον κύριο Νόισερ για την θετική του συνεισφορά. Σημαντική έκθεση για δύο λόγους. Πρώτο, οι διεθνείς διαπραγματεύσεις για την ε, αλλαγή του κλίματος έχουν, βρίσκονται σε εξέλιξη και επομένως για τους επόμενους στόχους θα είναι στο Παρίσι και 2015 πρέπει ε, να έχει κάτι να, να πει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα η συμβολή του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Πράσινη Βίβλο έχει τεράστια σημασία, διότι τον επόμενο Μάρτιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει το θέμα αυτό στην βάση προτάσεως της Κομισιόν. Ο δε πρόεδρος Μπαρόσο περιέλαβε στον λόγο του State of the Union το ότι μέχρι τέλους του έτους η Κομισιόν θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις. Δεύτερος λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό και για την για την εγχώρια προοπτική, μιλούμε για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, είπε ο κύριος ε, Νόισερ και για την διασυνοριακή ε, κίνηση της ενέργειας. Αυτό χρειάζεται μακροπρόθεσμη προοπτική. Γι' αυτό το λόγο θεωρεί η Κομισιόν ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό και ευχαριστούμε την ε, Επιτροπή Αναπτύξεως η οποία συμβάλλει με τον τρόπο αυτό στη μελέτη του θέματος. Ευχαριστώ. Κύριε αν έχετε πάρει το λόγο για να εξαγάγετε τελικά συμπεράσματα. Μετά από τα συγχαρητήρια της Προέδρου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν έχω τίποτε άλλο να προσθέσω. Merci. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία καταθέσεων τροπολογιών λύγει στις 15 Οκτωβρίου το μεσημέρι. Μου μένει μόνο, να ρωτήσω βέβαια αν υπάρχουν διάφορα, και αλλιώς να σας ανακοινώσω την ημερομηνία της επόμενης συνεδριάσεώς μας που θα είναι Δευτέρα 4 Νοεμβρίου στις 3 το απόγευμα και η επόμενη μέρα, ε, Τρίτη 5 Νοεμβρίου, τις συνήθεις ώρες του πρωινού και του απογεύματος. Σας ευχαριστώ όλες και όλους και θα σας δω τον Νοέμβριο.